Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, λάβετε θέσεις, έχει θέσεις πίσω. Θα προεδρεύσω σήμερα και αύριο, γιατί η πρόεδρος είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και μετά τα πρακτικά. Στις 21 Οκτωβρίου εγκρίθηκε η αναθεωρημένη έκδοση των κατευθυντηρίων γραμμών που συμπεριλαμβάνουν τροπολογίες του Κοινοβουλίου. Καλωσορίζω τους εμπειρογνώμονες που δεν έχουν ακόμη έρθει, άρα δεν τους καλωσορίζω ακόμη. Θα τους καλωσορίσω όταν θα έρθουν. Θα υπάρχει αναμετάδοση από το Web Stream. Με μεγάλη ευχαρίστηση τώρα θα οργανώσουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βρούνο Κοκέ, πρόεδρο της ΕΜΚΟ για τις πολιτικές απασχόλησης στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης και της θερατικής Ευρώπη 2020. Φυσικά θα τεθούν και ερωτήματα μετά την παρουσίαση όμως. Α, χαίρετε, εγώ θα μιλήσω γαλλικά, αν δεν απατώμε. Θα χωρίσω την παρουσίασή μου σε δύο τμήματα, γιατί περιλαμβάνει δύο θέματα. Πρώτον, η διακυβέρνηση, η διαχείριση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και μετά κατάσταση της αγοράς, εργασίας, της αγοράς εργασίας και μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης αυτήν. Για τη διαχείριση της στρατηγικής 2020, governance όπως λέμε, ε, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ έγινε την περασμένη εβδομάδα και είχαμε προετοιμάσει σχέδια συμπερασμάτων που εγκρίθηκαν και που ανταποκρίνονται στην εντολή που είχε αναλάβει το Συμβούλιο από τον Ιούλιο και που συνίστατο στην αναζήτηση μιας διαδικασίας ελαφρότερης, ελαφρύτερης και αποτελεσματικότερης ώστε το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ να μπορεί να έχει περισσότερα αποτελέσματα γενικά στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πολιτική της απασχόλησης. Η απάντηση που δώσαμε στην ΕΠΣΚΟ στην παραγγελία αυτή ήταν πρώτον βασιζόταν στα εξάμεινα των Προεδριών και το πρώτο από αυτά κατέληγε, θα κατέληγε στις αρχές Ιανουαρίου σε, μία, σε έναν απολογισμό της αγοράς εργασίας και περιγραφή όλων των πολιτικών προγραμμάτων και μετά η Αρινή Σύνοδος θα καθόριζε τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων τέλος έγκριση των συστάσεων τον Ιούλιο προς συγκεκριμένες χώρες. πρώτη συμβολή της ΕΠΣΚΟ σε αυτό το εξάμεινο θα συνίσταται με βάση τις δημοσιεύσεις της Κομισιόν σε χορήγηση ορισμένων συγκεκριμένων μηνυμάτων για τη στρατηγική που πρέπει να εγκριθεί για την πολιτική της απασχόλησης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της πολέμηση της ανέχειας, όλα αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Και η δεύτερη φάση στην οποία θα αντιδράσει η ΕΠΣΚΟ είναι μετά την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων τον Απρίλιο για τις μεταρρυθμίσεις, το ΕΠΣΚΟ θα εξετάσει και θα εγκρίνει τις συστάσεις προς τα κράτη-μέλη με βάση τις προτεραιότητες που θα έχει καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και των απαντήσεων που θα έχουν δώσει τα κράτη-μέλη ως εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Και μετά οι συστάσεις αυτές θα εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουλίου. Και τρίτη φάση την οποία παρεμβαίνει η ΕΠΣΚΟ δεν είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου όπως το καθόρισε η Κομισιόν, είναι πιο άτυπο, κάτι πιο ανεπίσημο, στα τέλη του έτους. Διότι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο όπως έχει καθοριστεί είναι για λήψη αποφάσεων, αλλά δεν προβλέπει καμία φάση αποτίμησης, αξιολόγησης, γνωστοποίησης, επιτήρησης του τι συμβαίνει στα διάφορα κράτη-μέλη και ως προς τη συγκυρία της αγοράς εργασίας και ως προς τη δομική πτυχή. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το δεύτερο εξάμεινο πρέπει να αφιερωθεί στη συλλογή στοιχείων αποτίμησης, αξιολόγησης, διάγνωσης και ανταλλαγής πληροφοριών για το τι συγκεκριμένα συμβαίνει στις χώρες μέλη. Είπαμε λοιπόν στο τέλος του χρόνου το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ να πληροφορηθεί από την ΕΜΚΟ, από την Κομισιόν και από όλους τους ενδιαφερόμενους που θα το ήθελαν για το ποια είναι η κατάσταση των μεταρρυθμίσεων στις διάφορες χώρες. Αυτό βέβαια δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί γιατί φέτος υπάρχουν προπρογράμματα εθνικών μεταρρυθμίσεων, προσχέδια προγραμμάτων και θα δούμε τι λένε αυτά τα σχέδια και μετά θα δούμε ποιες προτεραιότητες προκύπτουν από τις χώρες μέλη. Αλλά το 11 θα αλλάξουν τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε αυτά τα, αυτές τις τρεις φάσεις, δύο επίσημες, αντίδραση στις προτάσεις Κομισιόν για γενικές κατευθυντήριες γραμμές στην Αρνή Σύνοδο συστάσεις προς τα κράτη-μέλη ως προς τις προτεραιότητες τους για τις μεταρρυθμίσεις τον Ιούλιο και τρίτη φάση της διαχείρισης ΕΠΣΚΟ η αξιολόγηση των τεκτενομένων στα κράτη-μέλη στα τέλη του χρόνου. Και μετά θα αρχίσει νέος άλλος κύκλος με καινούριο ευρωπαϊκά εξάμεινα. Αυτά λοιπόν προτείναμε εμεί και τα δέχτηκε και το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ την περασμένη εβδομάδα. Δεύτερον, η οικονομική κατάσταση και ιδιαίτερα της αγοράς εργασίας και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την καταπολέμηση της κρίσης. Εδώ μαζί με την Κομισιόν είχαμε συγγράψει ένα έγγραφο ως βάση μια συζήτησης στα γεύματα της ΕΠΣΚΟ. Γενικά το έγγραφο αυτό κάνει μια γενική αξιολόγηση του τι έγινε από την κρίση και μετά αύξηση της ανεργίας που έπληξε ιδιαίτερα τους μισθωτούς, τους πιο ευάλωτους με πρόθεσμα συμβόλαια, τους νέους και τα λοιπά. Νομίζω τα γνωρίζετε ήδη αυτά. Σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση σταθεροποιήθηκε στην αγορά εργασίας, η ανεργία σταμάτησε να αυξάνεται στο σύνολο της Ένωσης, η απασχόληση επίσης σταθεροποιήθηκε. Ε, Mais bon, euh, rien de... Και τελικά δεν πρόκειται ακόμη για αναθέρμανση, μόνο για σταθεροποίηση. Λοιπόν, είναι ακόμη δύσκολα λοιπόν τα πράγματα και πρέπει να προσθέσουμε ότι η κατάσταση στις διάφορες χώρες μέλη παραμένει εξαιρετικά ετερογενής, αντίθετα από προηγούμενες πιο ήσυχες περιόδους ανάπτυξης ή και υπαναχώρησης υπήρχε μια ομογένεια, ενώ εδώ τώρα υπάρχει τεράστια ετερογένεια. Στην τελευταία μηνιαία έκθεση της Κομισιόν για την Αγορά Εργασίας τον Οκτώβριο την περσμένη εβδομάδα υπάρχουν πίνακες που δείχνουν ότι υπάρχει αυτή η ετερογένεια σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό σημαίνει ότι πέρα από τη σταθεροποίηση αν εξετάσουμε τις χώρες μία-μία βλέπουμε ότι η κατάσταση διαφέρει πάρα πολύ από τη μία στην άλλη και δεν υπάρχει κοινή συνταγή για όλους, ακόμη λιγότερο από ό,τι πριν. Αυτό είναι πραγματική δυσκολία και τρίτον δεν ξέρουμε καθόλου ποια είναι η σχέση μεταξύ ανάπτυξης και απασχόλησης. Για οποιαδήποτε χώρα δεν το ξέρουμε αυτό γενικά. Εγώ είμαι οικονομολόγος και θα μπορούσα να σας πω ότι δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Βέβαια δίνονται τοπικές εξηγήσει ότι στη Γερμανία υπάρχει μερική ανεργία σε σύγκριση με άλλες χώρες κτλ. Αλλά γενικά η σύνδεση, η σχέση ανάπτυξης και απασχόλησης δεν είναι σαφής και είναι πολύ δύσκολο να δώσει κανείς μια οδηγία κοινή για όλους. Μπορούμε όμως να δούμε τι αντιμετωπίστηκε επιτυχώς. Τα μέτρα μερικής ανεργίας που εφάρμοσαν οι περισσότερες χώρες, όλες όσες τα εφάρμοσαν ικανοποιήθηκαν. Αν και μερικές φορές ε, στήχησε πολύ. Μετά υπήρξαν τα προγράμματα ενεργοποίησης λέει ο μιλητής. Μετά από τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης υπήρξαν τα προγράμματα ενεργοποίησης των ανέργων που ήταν πιο αποτελεσματικά όταν στόχευαν συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, τους νέους, ας πούμε, κλπ. Τα προγράμματα αυτά ενεργοποίησης ε, είχαν αποτέλεσμα. Και τρίτο είδος πολιτικής που εφαρμόστηκε εκπαίδευσης ή μετεκπαίδευσης διότι κατάρτισης γιατί επειδή υπήρχαν πολλοί άνεργοι πολλές χώρες μέλη θέλησαν να εφαρμόσουν τέτοια προγράμματα κατάρτισης και όταν συσχετίστηκαν με τα μέτρα σχετικής ημερικής ανεργίας δεν δούλεψαν. Αντίθετα, πολλοί άνεργοι ή μισθωτοί είχαν αποτέλεσμα από τα προγράμματα αυτά κάθε αυτά. Και τέλος, η ελάφρυνση των κοινωνικών εισφορών οδήγησε στη δημιουργία ορισμένων περισσότερων θέσεων εργασίας παντού και η μέθοδος αυτή συνεχίζει να εφαρμόζεται ως αντιμετώπιση της κρίσης. Διότι αυτό χρειάζεται τώρα, η έξοδος από την κρίση, αφού σταθεροποιήθηκε η αγορά εργασίας. Αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν και οι περικοπές των προϋπολογισμών που μας υποχρεώνουν να καθορίσουμε προτεραιότητες στην πολιτική της απασχόλησης. Αυτό το θέμα είχε θέσει η Βελγική Προεδρία κατά το γεύμα της ΕΠΣΚΟ με βάση το έγγραφό μας και το θέμα αυτό λοιπόν ήταν ποια προτεραιότητα έχετε στον προϋπολογισμό σας και τι πολιτική θα διατηρήσετε έναντι των υπολείπων σε αυτήν τη φάση της ανάκαμψης που δεν υπάρχει. Τα προγράμματα που επέλεξαν τα κράτη-μέλη με βάση αυτά που είπαν οι υπουργοί κατά τα δύο τρίτα ανέφεραν το θέμα των νέων γιατί η ανεργία των νέων αυξήθηκε πολύ, το ξέρατε αυτό ήδη και οι προπολογισμοί γενικά διατηρούν τα προγράμματα για την υποβοήθηση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας κτλ. Δεύτερο είδος μέτρων που δέχτηκαν τα κράτη-μέλη η ελάφρυνση των κοινωνικών εισφορών για τις νέες θέσεις εργασίας. Εδώ καταλαβαίνουμε εύκολα γιατί, γιατί από προοπτική δημιουργείται μια θέση εργασίας, δεν τις αφαιρούμε εισφορές και έτσι δημιουργούμε περισσότερους πόρους για το δημόσιο προϋπολογισμό. Τρίτο είδος μέτρων που επέλεξαν τα κράτη-μέλη η μεταρρύθμιση, για να το πω έτσι, των εισφορών ανεργίας, των επιδομάτων ανεργίας. Ενώ αναπτυσσόταν η κρίση, πολλές χώρες μείωσαν τα κριτήρια εκλογιμότητος ώστε να μπορεί κανείς πιο εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτά τα επιδόματα και αύξησαν και τις περιόδους αποζημίωσης. Στη φάση της ανάκαμψης όμως δεν αποφάσισαν να το συνεχίσουν, να καταργηθούν τα έκτακτα μέτρα και να υπάρξει μεγαλύτερη λιτότητα στο σύστημα των αποζημιώσεων ενέργειας, επιδομάτων ενέργειας, ώστε να γίνουν όλα αυτά πιο στοχευμένα. Τρεις λοιπόν οι προτεραιότητες. Οι νέοι, η ελάφρυνση των κοινωνικών εισφορών στις νέες θέσεις και μεταρρύθμιση των επιδομάτων ενεργείας. Επίσης νομίζω ότι πολλοί μίλησαν για συγχρηματοδότηση, δηλαδή για πολλά από αυτά τα μέτρα αναζήτησαν τα κράτη εταίρους. Ευρωπαϊκά ταμεία, κοινότητες, να υπάρξει ένα μοίρασμα δηλαδή του βάρους και μεγάλος αριθμός υπουργών είπε επίσης ότι ο προϋπολογισμός της χώρας τους ε, μεταφέρθηκε κατά μεγάλο βαθμό στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι πλήρως βέβαια, όχι, όχι καθόλου. Θα μπορούσε, αν και δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες των μέτρων αυτών, αλλά γενικά στην κοινωνική πολιτική και στην πολιτική απασχόληση απασχόλησης είπαν ότι το τοπικό επίπεδο μπορεί να ανταποκριθεί καταλληλότερα εφόσον μάλιστα υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά από περιφέρεια σε περιφέρεια και ότι επομένως οι υπουργοί και οι χώρες το σκέφτονται όλο και σοβαρότερα. Εκτός από αυτά, στο έγγραφό μας, στο οποίο βασίστηκε η συζήτηση, επιλέξαμε με την Κομισιόν να τονίσουμε ιδιαίτερα τρεις μεθόδους για την αναθέρμανση. η αναγκαιότητα να δούμε πώς θα βγούμε από τα μέτρα, όχι καταργήσουμε, πώς θα βγούμε από τα μέτρα αυτά μερικής ανεργίας, δηλαδή να διατηρηθούν τα μέτρα, όχι να καταργηθούν αμέσως, αλλά ή και καθόλου ποτέ, αλλά να δούμε πώς θα περιοριστεί ο προπολογισμός τους, γιατί στρεβλώνει κάπως την αγορά. Δεύτερη προτεραιότηση. η αναγκαιότητα να ενδυναμωθούν τα στοχευμένα και ενεργά μέτρα για απασχόληση, λίγο όπως λένε οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, από εδώ και πολύ καιρό που επαναλάβαμε και εμείς, και τρίτον, μια προσπάθεια, να γίνει μια προσπάθεια καλύτερης εξέτασης των διατάξεων της ασφάλισης ανεργίας όπου μπορούν να γίνουν μάλλον και εξοικονομήσεις και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να προστατεύονται καλύτερα οι μισθωτοί. Αυτά. Και αν έχετε απορίες, ευχαριστώ να τη λύσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Κύριε Σεσέρκους, πρώτο στο κατάλογο. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας έδωσε η Βελική Προεδρία. Με λεπτομέρειες και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό γιατί τελευταία οι άνεμοι που φυσούν από το Συμβούλιο περιλαμβάνουν μια τακτική έτσι λύθη του Κοινοβουλίου και του ρόλου του. Και αυτό είναι κάτι τακτικό και διαρθρωτικό. Δεν είναι κάτι το περιστασιακό. Σα ευχαριστώ πολύ για τι πληροφορίε, τι διαρθρωμένε και λεπτομέρειε που μα δώσατε και που αφορούν αυτή την ε, δύσκολη στιγμή για την απασχόληση στην ε, Ευρώπη. Το μόνο πρόβλημα, κύριε Κοκέ, είναι το ότι δεν ξέρω ακριβώς αν το θέμα της διακυβέρνησης αν αντιμετωπίζεται εκεί που πρέπει, στο κατάλληλο μέρος. Δεν ξέρω αν είναι στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, το συμβούλιο το οποίο ανησυχεί για την κρίση της απασχόλησης, για την κρίση γενικότερα, φαίνεται ότι ξεχνάει το θέμα αυτό της απασχόλησης. Όπως είδαμε στην task force του κ. Βαντρομπά την μελλοντική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Αυτό είναι μια υποψία που έχω, ίσως κάτι παραπάνω από υποψία, ότι πολλές φορές λέμε πολλά λόγια τη στιγμή που το σχήμα της πραγματικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης βρίσκεται αποκλειστικά όχι μόνο επικεντρωμένο στα οικονομικά ζητήματα, αλλά λεπτομερέστερα στα θέματα τα φορολογικά, ούτε καν στην ανάπτυξη. Και εσείς λέγατε σωστά ότι διάφοροι παράγοντες δεν ε, συμφωνούν σχετικά με την ε, σχέση που υπάρχει μεταξύ απασχόλησης και ανάπτυξης. Υπάρχει όμως νομίζω μια βασική ομοφωνία όσον αφορά το δόγμα που λέει ότι ο, αν ασχοληθούμε μόνο με την ε, φορολογική μεταρρύθμιση σκοτώνοντας τα προγράμματα δηλαδή τα οποία θα μπορούσαν να οδηγούν σε μια αύξηση της ζήτηση, σε αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κτλ. τότε αυτό θα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις για την απασχόληση. Εγώ δυστυχώς βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης και την ταχεία έξοδα από την κρίση. Για, για όλες τις χώρες ισχύει το ίδιο είτε για αυτές που πρέπει από το 12 να πάνε στο 3, είτε από αυτές που πρέπει να πάνε από το 6 στο 3. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι η ίδια. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά η ΕΣΚΟ να μας δώσει ουσιώδεις ρεαλιστικές απαντήσεις που αντανακλούν την πραγματικότητα στην κάθε χώρα. Βλέπω όμως ότι και πάλι όσον αφορά την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση μας δράβουν ένα κουστούμι που θα το φορέσουν όλοι και το οποίο θα είναι πολύ στενό για πολλούς. Και νομίζω ότι δυστυχώς αυτό θα αυξήσει, δεν θα λύσει τα προβλήματα. Οπότε κύριε Κοκέδη ρωτώ με το εξή. Το Συμβούλιο, το ΕΠΣΚΟ, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορούσε πριν η προχωρήσει η task force του κ. Φαντρομπάη μήπως εσείς θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι σε σχέση με την κοινωνική διάσταση της κρίσης. Μήπως εσείς θα μπορούσατε να συμφωνήσετε και με το Κοινοβούλιο και με πολλούς άλλους οι οποίοι λένε ότι δεν είναι αυτή η λύση που θα βγάλει την Ευρώπη από την κρίση της απασχόλησης. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι το εξή. Είχα μια προσωπική εμπειρία αυτό το Σαββατοκύριακο. Βλέπω ότι εσείς στο Συμβούλιο, όπως και στο Κοινοβούλιο, ανησυχούμε τόσο πολύ με το θέμα της μαζικής ανεργίας των εκατομμυρίων Ευρωπαίων που έχασαν την δουλειά τους και αναζητούν δουλειά και ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει πολύ δουλειά σε σχέση με την υγεία, με την ποιότητα της απασχόλησης και ταυτόχρονα βλέπουμε να διαβρώνονται και άλλα συστατικά σημαντικά όπως η ποιότητα της εργασίας και έχουμε εγκαταλείψει παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί νομίζω δεν θα πρέπει μόνο να ασχολούμαστε με την ποσότητα της απασχόλησης αλλά και την ποιότητα της απασχόλησης μπροστά σε αυτό το δράμα, σε αυτή την καταιγίδα που αφορά την απασχόληση και που είναι κάτι το δραματικό. Γι' αυτό ακριβώς ρωτάω, το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα μας συνοδεύσει θα συμπορευτεί μαζί μας στο να δώσουμε έμφαση στα θέματα της ποιότητας απασχόλησης που ταλανίζουν σήμερα εκατομμύρια Ευρωπαίων λόγω ακριβώς της κακής ποιότητας απασχόλησης που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Τόμας Μάν. Ε, Σας ευχαριστώ. Αναφέρατε κύριε ότι έχουμε ένα στάδιο σταθεροποίησης χωρίς να έχουμε ανάκαμψη. Βέβαια, είναι σωστό. Σταθεροποίηση είναι σημαντική καταρχήν για να μην περάσουμε σε μια εφορία που να μας οδηγήσει στο να κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Βλέπω επίσης ότι πολλοί στη Γερμανία παραδείγματος χάρη ό,τι θετικό στοιχείο υπάρχουν στον εξωτερικό τομέα ε, δεν φτάνει μέχρι τον κάθε πολίτη. Δεν έχει την εντύπωση ότι πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν, πολύ μακριά είμαστε. Δεν κατανοούν ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία. Πρέπει πολλά να γίνουν, σαφώ, αλλά αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εάν όλοι οι πολίτε έχουν την εντύπωση ότι καταρχήν μπορούμε να συμμετάσχουμε, έχουμε δυνατότητε, γινόμαστε πιο καλά αποδεκτοί, αηφόρα και μακροπρόθεσμα. Δεύτερον, γιατί είναι τόσο δύσκολο στα διάφορα κράτη-μέλη εκείνοι που έχουν την ευθύνη να πούνε ότι θα πρέπει να προωθήσουμε περαιτέρω μεταρρυθμίσει. Γιατί λέμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε τα χρήματα που έχουμε, να οδηγηθούμε σε παγίωση, να πούμε ότι θα πρέπει σωστά να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά μας, να μην πούμε ότι έρχονται τώρα οι καλοί καιροί και μπορούμε να έχουμε πολλές απαιτήσει και να επενδύσουμε όπως θέλουμε. Λέγεται όμως ότι μας τροχοπεδείται πολύ ισχυρά, όπως είπε και ο κύριος ε, Τσέρκας προηγουμένως. Το θέμα της ε, ανεργίας ε, στο παρελθόν ε, είχαν πάρει επιχειρήσεις επιδοτήσεις από το κράτος για να μην χάσουν τις θέσεις απασχόλησης που είχαν. Χρησιμοποίησαμε δηλαδή φορολογικά έσοδα, ούτως ώστε να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, ούτως τόσο που περνάμε σε μια καλύτερη φάση, να τους πούμε ναι, εδώ είσαστε, δεν έχετε περάσει από τη μάστιγα αυτή της ανεργίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εσείς πώς, ε, τι, τι, τι μέλλον θεωρείτε ότι θα έχουν αυτά τα μέτρα σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί τώρα ζητούν εργαζόμενους, δεν μπορούμε όμως κάνουν μεγάλες εταιρείε να πούνε ότι ας έρθουν από όλο τον κόσμο που τους βρούμε. Όχι, να πούμε εκείνοι που είναι εδώ, εκείνοι που ξέρουμε πώς εργάζονται, να προσληφθούν. Να τους πούμε εδώ είσαστε, εσάς θέλουμε. Τελευταία παρατήρηση. Ο Σάλφος Έρκας ε, αναφέρθηκε στο σύμφωνο σταθερότητα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε έχουμε το σύμφωνο σταθερότητας και κάποιους αυτοματισμούς και τα πάντα θα πρέπει να ισχύουν για όλους. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται κάστοτε. Να πούμε στα κράτη-μέλη θα πρέπει να μελετήσετε τα πράγματα όπως πρέπει. Όχι επειδή τρεις-τέσσερις χώρες θέλουν αυτοματισμό, αλλά να μπορέσετε να συμμετάσχετε όλοι για να μπορέσουμε από κοινού να διαπτώσουμε μια στρατηγική αηφορίας. Αν θέλουμε να αποχαιρετήσουμε το σύμφωνο σταθερότητα δεν αξίζουν τίποτα αυτά που έχουμε κάνει από κοινού. Να δούμε δηλαδή ότι θα πρέπει πραγματικά η στρατηγική αηφορία να είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και σα ρωτάω τώρα, θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πλειοψηφία ή θα πρέπει να ασχολούμεθα ψυχνά ακριβώ ε, στι συνεδριάσει των Υπουργών Οικονομικών να ακούμε κάποιε ε, δηλώσεις για τι οποίε εμεί να λέμε ότι αυτά θα τα περιμέναμε. Ε, τι αγοραπολισίε είναι αυτέ. Ε? εγώ είμαι κατά του να υπάρχει αυτή, αυτού του τύπου συνέλεγη. Ευχαριστώ, κυρία Τόρνα. Yes, um, thank you for... Να ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχω μια ερώτηση σε σχέση με αυτά που είπατε για μια νέα task force της ΕΠΣΚΟ που θα τροφοδοτεί τις συζητήσεις που γίνονται για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Πολύ θετική αυτή η προοπτική, όμως έχω μια ερώτηση. Θα ήθελα την άποψή σας σχετικά με τη νέα οικονομική διακυβέρνηση όπως αυτή παρουσιάστηκε από την Κομισιόν στα τέλη του Σεπτέμβρη όπου δεν είδα να υπάρχει καμία αναφορά στην απασχόληση ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στην κάθε χώρα μέλος. Έγινε λόγος περισσότερο για την οικονομική ανάπτυξη και τα συστήματα κυρώσεων. Δεν είδα καμία αναφορά λοιπόν στην μεταρρύθμιση του 2005, δηλαδή στο Σύμφωνο Σταθερότητας, όπου για πρώτη φορά αφαιρέθηκε η απασχόληση ως ένα βαρύδι, κάτι το οποίο θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας όταν εμείς αλλάζαμε τις οικονομικές πολιτικές μας. Πώς ε, βλέπετε εσείς λοιπόν αυτό το σχέδιο της Κομισιόν για την οικονομική διακυβέρνηση γιατί δεν βλέπω να υπάρχει η απασχόληση που είναι ακρογωνία λίθος του όλου συστήματος και λυπάμαι γι' αυτό. Και βλέπω ότι το ΕΠΣΚΟ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και βλέπω να υπάρχουν έτσι αποκλίνουσες τάσεις. Ποια είναι η απόψη σας από αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ελίζα Μπεσσιραντέρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Και ιδίω να διαβάσει τα συμπεράσματα, είδα ότι υιοθετήσετε πολλά από τα συμπεράσματα του Κοινοβουλίου και σας συγχαίρω. Πραγματικά μπορώ να πω ότι η Βελική Προεδρία συνεργάζεται ασυνήθιστα καλά, θα έλεγα, με το Κοινοβούλιο. Πολύ ασυνήθιστα. Και ιδίω αυτά που αποφασίζουμε για την έκθεση Jobs τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης είναι εδώ, στη δική σας παρουσίαση, πολύ καλό αυτό, και μας είπατε και ποια θα είναι η συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί και ο έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καλά ακούγονται όλα αυτά, έχω αμφιβολίες κατά πώς θα πετύχουν. Γιατί αν δεν υπάρχει ενθουσιασμό στα κράτη-μέλη να τα εφαιρήσουν αυτά, μπορείτε εσείς ε, τυπικά να προωθήσετε τις διαδικασίες αυτές, αλλά δεν θα πετύχετε πραγματικά τροποποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει ενθουσιασμό αυτό. Και ιδίω όσον αφορά τι πράσινε θέσει εργασία και το θέμα των νέων ικανοτήτων για νέες θέσει απασχόληση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στα συμπεράσματά σα, δεν ξέρω, υιοθετώντα αυτή την πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου, μπορείτε πραγματικά να δώσετε μια όθηση για να υπάρχει αυτό ο ενθουσιασμό στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μα πείτε κάτι σχετικά. Ευχαριστώ κύριε Στάινπρο. Ähm, Ορισμένοι από τους σε αναφέραν αυτό που θέλω να φέρω κι εγώ. Εξ στον ομάδα μας θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ορισμένες από τις ιδέες της Επιτροπής αυτής περνάνε στις ε, κατευθύνες γραμμές για την πολιτική απασχόληση, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν και μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία, καλύτερη μάλιστα συνεργασία από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό για το μέλλον θα μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη πιο θετικά. Γιατί υπήρχαν ορισμένε προσθήκε που για τη δική μα επιτροπή εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Και θα ήθελα να σα παρακαλέσω να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω στα θέματα αυτά που είναι τόσο σημαντικά για μας εδώ στο Κοινοβούλιο και ίσως ας πούμε αυτά τα θέματα παραδείγματος οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν δυσκολία να ενσωματωθούν στην αγορά απασχόλησης αυτές οι ομάδες να προωθούνται περισσότερο και στο μέλλον ελπίζω να έχουμε την υποστήριξή σας εδώ και δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε κά ποια πράγματα που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε στο μέλλον. Αυτά κατά τα άλλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ κύριε Βαλτασάρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βεβαίω και εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για την παρουσίαση του κυρίου Κοκέ. Και νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις για την σταθερότητα που φαίνεται ότι πετυχαίνουμε σιγά σιγά βγαίνοντας από την κρίση φαίνεται ότι αντιβαίνουν σε κάποια στοιχεία, σε κάποια δεδομένα. Δηλαδή κάποιες χώρες μέλη έχουν φτάσει σε μεγάλα επίπεδα εξαγωγών, η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μου έφτασε στα επίπεδα του 95, όμως όλα αυτά δεν λύνουν ποδενή το θέμα της απασχόλησης. Δηλαδή αυτά που χάθηκαν παραμένουν ως απώλεια. Δηλαδή χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας έχουν χαθεί και δεν έχουν ανακτηθεί. Αυτή λοιπόν η αύξηση της ε, βιομηχανικής παραγωγής δεν ανακτά τις χαμένες θέσεις εργασίας. Και μάλιστα στις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης προστίθενται προβλήματα τα οποία ήταν παρόντα παλαιότερα και που συνεχίζουν να είναι παρόντα. Δηλαδή η δυσκολία που αντιμετωπίζει όλος ο μεταποιητικό τομέας στην Ευρώπη, ο ανταγωνισμός από τις αναπτυσσόμενες χώρες οδηγεί στην ε, μετακόμιση παραδοσιακών βιομηχανιών και επιχειρήσεων που φτιάχνουν μάλιστα και παραδοσιακά προϊόντα. Πρόσφατα είχαμε το περιβόητο παράδειγμα μιας εταιρείας που έφτιαχνε τσάι αγγλικής και που θα παράγει εκτός Ευρώπης. Το πρόβλημα λοιπόν που τίθεται και που κάποιο και εδώ προσπάθησε να αντιμετωπίσει είναι το κατά πόσο η Ευρώπη θα μπορούσε να συνεχίσει να έχει ακόμα ένα, ευρωπαϊκό σύστημα, ένα βιομηχανικό σύστημα ή κατά πόσο εμεί θα είμαστε οι παραλήπτε τμήματων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κτλ. που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου σε εμά. Οπότε εδώ έχουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, καταπολέμηση της στόχιας, έλλειψη απασχόλησης και τα λοιπά, τα οποία φαίνεται ότι δεν έχουμε εργαλεία για, να πολεμήσουμε ως φαινόμενο. Και ενώ υπάρχουν νέοι τομείς ε, οικονομικοί όπου επεκτείνεται η οικονομία, οι δυνατότητες απορρόφησης θέσεων εργασίας είναι περιορισμένοι όσον αφορά δηλαδή την απώλεια θέσεων εργασίας που έχουμε και την, ε, το αίτημα για θέσεις εργασίας που ζητάει νέα γενιά. Όλα αυτά κάνουν και τα σύμφωνα σταθερότητα ακόμα πιο αυστηρά. Γνωρίζουμε λοιπόν αυτή την αντίφαση και θεωρούμε ότι η δημιουργική και η πολιτιστική βιομηχανία αποτελεί μια προοπτική για το μέλλον. Όμω οι χώρε μέλη περικόπτουν όλε τι χρηματοδοτήσει του πολιτισμού. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ανάπτυξη και μεγέθυνση για τις επιχειρήσεις, όμως τα σύμφωνα σταθερότητας μειώνουν και τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων που ως Ευρωπαϊκή Ένωση προορίζουμε στους στόχους του, της ε, κατηγορίας 1 για τη συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω κάνει δύσκολη, εάν δεν αποκλείει τελείως, τους ε, τομείς μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισης όπου θα έχουμε ζημιές κοινωνικές που είναι δύσκολο να διορθωθούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι παρά τα πρώτα δείγματα δεν έχουμε ακόμα κάποια ιδέα για το τι γίνεται στις χώρες μέλη. Και δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι γίνεται, δεν είναι ακόμα σαφές ποιοι είναι οι στόχοι και ποιες θα είναι οι επιλογές οι οποίες όχι μόνο θα μας βγάλουν έξω από την κρίση αλλά θα μας οδηγήσουν στο να ανακτήσουμε όλη αυτή αυτή την δέσμη της απασχόλησης που έχουμε χάσει. Διαφορετικά θα πρέπει από το και στο εξή να λέμε ότι το 20% των, ε, της ανεργίας στην Ευρώπη είναι αυσιολογικό και θα πρέπει να το διατηρήσουμε με το κοινωνικό κράτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντέρη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι είναι πια καιρός να βγούμε από την κρίση. σας βρίσκω πολύ αισιόδοξο και αυτό είναι θετικό. Αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Επίσης μιλήσατε για την κατάρτιση. Θα ήθελα να μου πείτε μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τις κλιματολογικές αλλαγές. Και όπως είπε και η συνάδελφος Ελισάβετ Σρότερ, Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, τι συνοδευτικά μέτρα προβλέπετε. Μιλήσατε για κατάρτιση. Θέλω λοιπόν να μάθω με ποια, εργα... ποια εργαλεία θα δώσετε στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν αυτές τις νέες προκλήσεις ώστε οι μισθωτοί να έχουν την κοινωνική τους ασφάλιση Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Σε περίοδους κρίσης, βλέπουμε τι γίνεται και στη Γερμανία, δεν απολύουν αλλά κάνουν μια κατανομή της εργασίας, δηλαδή στο χρόνο εργασίας. Δεν είναι καιρό να αναρωτηθούμε και γι' αυτό, για την κατανομή της εργασίας, να δουλεύουν όλοι λιγότερο για να δουλεύουν περισσότεροι. Τρίτο ερώτημα εφόσον υπάρχει κρίση της απασχόλησης, βλέπουμε ότι υπάρχουν δυστυχώς δύο τομείς οι μισθωτοί που είναι τα μεγαλύτερα θύματα και οι πρόεδροι των επιχειρήσεων που έχουν πριν. Πότε λοιπόν θα εφαρμόσουμε επιτέλους μία σοβαρή κοινωνική δημοκρατία στις επιχειρήσεις. Αυτή την ιδέα τη συζήτησε καθόλου το Συμβούλιο. Τέλος για τους νέους και τις νέες. Αυτοί και αυτές περιμένουν πολλά από την Ευρώπη κύριε Πρόεδρε μου. Και όλο και περισσότερο στην καθημερινή του ζωή ακούνε να γίνεται λόγος για ανασφάλεια. Ποια εργαλεία λοιπόν προβλέπετε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτής της νεολαίας που δεν έχει λύσεις μπροστά της. Ευχαριστούμε πολύ. Φαίνεται από τη συζήτηση ότι το θέμα που τίθεται περισσότερο είναι πώς θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τη δουλειά σας με τη δική μας δηλαδή μετά τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών. Τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή Απασχόλησης. Μπορεί και εσείς να λάβετε υπόψη σας μερικές από τις απόψεις του Κοινοβούλιο ας πούμε. Για πολλά θέματα από αυτά που τέθηκαν όπως της κυρίας Σρότερ τέθηκε το θέμα αυτό της συνεργασίας αλλά συχνά βλέπουμε ότι στην Επιτροπή μας διαπιστώνουμε ότι η δουλειά μας τελικά δεν συνδέεται και πολύ με τη δική σας, ίσως θα έπρεπε. Ίσως να διαθέτετε ένα τέταρτο για τις απαντήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης Μπορεί να έρθει να σας μιλήσει όποτε θέλετε, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Τώρα πιο συγκεκριμένα πώς να γίνονται πιο επίσημα και τακτικά τέτοιες ε, ανταλλαγές απόψεων. Σας μίλησα για τις τρεις φάσεις, διαχείριση κλπ, όπως τις είχε εγκρίνει το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ την περασμένη εβδομάδα. Και η τρίτη, η λιγότερο επίσημη, αυτή που μιλάει για αξιολογήσεις ε, στο τέλος του έτους κτλ. Είναι νομίζω η καταλληλότερη για συνεννόηση και με το κοινοβούλιο για να ακουστούν νέες προτάσεις κλπ. Και όχι μόνο από το κοινοβούλιο αλλά και από τους κοινωνικούς εταίρους κλπ. Αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή. Μέχρι τώρα δεν ήταν ο καταλληλότερος χρόνος για να ακουστούν τέτοιες προτάσεις. Τώρα όμως είναι. Τώρα πιο επίσημα εγώ θα έλεγα ότι δυστυχώς μόνο τα σύντομα και εύληπτα μηνύματα ακούγονται. Αυτό σας το λέω έτσι ως συμβουλή γιατί εγώ μιλάω για την ΕΜΚΟ βέβαια, για το ετκο αλλά ναι. για την ΕΜΚΟ ακούμε από το Κοινοβούλιο πράγματα τα οποία αν είναι και τακτικά και σύντομα και εύληπτα δεν θα έχουμε πρόβλημα να τα συμπεριλάβουμε. Αν και επισήμως δεν μπορώ να σας κάνω καμία τέτοια υπόσχεση, το κατανοείτε εύκολα. Τώρα να προσπαθήσω να απαντήσω σε πέντε λεπτά σε όλες τις ερωτήσεις. Πρώτον, για τους περιορισμούς των προϋπολογισμών που είναι και το κυριότερο θέμα εδώ. Η Επιτροπή Απασχόλησης πρέπει, έχει καθήκον να εφαρμόζει πολιτικές, πολιτική ακριβώς απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας όπως τα επιδόματα ανεργίας ας πούμε και το θέμα εδώ είναι βεβαίως όπως είπε κάποιος από εσά, πόσο θα κρατήσουν όλα αυτά γιατί βραχυπρόθεσμα δεν υπάρχει επιλογή δεν έχουμε χρήματα και τα περισσότερα κράτη-μέλη λένε ότι έχουν πολύ περιορισμένους πόρους για τέτοιες αποζημιώσεις και άρα πρέπει να επιλέξουμε ό,τι έχει τον καλύτερο λόγο κόστος αποδοτικότητας. Έτσι ώστε να οδηγηθούν οι άνεργοι προς την απασχόληση, να έχουν βραχυπρόθεσμα κάποιο μήνυμο μισόδημα, με στόχο όμως να φτάσουν στην απασχόληση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και το θέμα είναι ότι είναι πολύ απειλητικό το πρόβλημα αυτό γιατί πολλά κράτη-μέλη αν δεν εφαρμόσουν τέτοια μέτρα θα καταστραφεί λίγο πολύ ολόκληρο το κοινωνικό του σύστημα προστασίας. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Ακόμη και αν δεν είναι εκεί το κύριο θέμα των εργασιών μας, αλλά το λαμβάνουμε δεόντως υπόψη. Τώρα, για να είναι βιώσιμα όλα αυτά πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη. Και το πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη προς το παρόν είναι αδύναμη ή όπως λέει η Κομισιόν δεν είναι δυνατή. Προς στιγμή τέλος πάντων δεν μπορούμε να προβλέψουμε κανένα ρόδινο μέλλον ως προς τον αριθμό της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ως προς τη χρηματοδότηση της πολιτικής κοινωνικής προστασίας και απασχολησιμότητας. Αυτό τι σημαίνει ότι, ότι λέγω, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές, ας το πω έτσι. Και οι μεγάλες αυτές αλλαγές πρέπει να αφορούν καταρχήν τη σφαίρα όπου δημιουργείται ο πλούτος, γιατί εκεί δημιουργούνται οι θέσεις απασχόλησης. Και εδώ είναι ο κόμπος. Αν δεν υπάρχει ανάπτυξη υπάρχει μείωση της δημιουργίας πλούτου και αυτό είναι αρνητικό για όλους. Οι περιορισμοί του προϋπολογισμού λοιπόν είναι ένα θέμα, άλλο όμως θέμα είναι η αναγκαιότητα να δημιουργηθεί ανάπτυξη και τρίτον ότι ένα από τα αρνητικά στοιχεία στον απολογισμό της Λισαβόνας είναι ότι δεν υπήρξαν προτάσεις μακροοικονομικές και μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας δεν συνδέθηκαν τα δύο αυτά θέματα. Ενώ ένας από τους στόχους της στρατηγικής που ζητούμε σήμερα είναι καλύτερο συνδυασμός τους. Έτσι νομίζω ότι απαντούμε στις ανησυχίες σας, ανταποκρινόμαστε. Το ΕΠΣΚΟ δεν μίλησε πολύ για τη διαχείριση όπως τη περιέγραψε η Κομισιόν το Σεπτέμβριο και αναρωτιέται κανείς αν το ΕΠΣΚΟ έχει ως προτεραιότητα την κοινωνική προστασία και την απασχόληση μέσα στα πλαίσια της νέας στρατηγικής. Σε αυτό θα απαντήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα, δεν θα απαντήσω εγώ, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι τα συμπεράσματα του ΕΠΣΚΟ δεν είναι ότι το εύκο βρίσκεται στο κέντρο του κόσμου, γράφεται μέσα σε μια ιστορία και στη στρατηγική που ενέκρινε υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία βασιζόμενα και στις ίδιες τις συνθήκες. Το θέμα όμως είναι αν θα ακουστεί, αν θα ακουστούν όλα αυτά. Και το ΕΠΣΚΟ αυτό ζήτησε ακριβώς. Να με ακούσει το Συμβούλιο αφού του δίνω τον νομική δυνατότητα διότι ακόμη κι αν η μακροπρόθεσμη πολιτική μακροοικονομική πολιτική δεν προβλέπει τίποτα ειδικά για την απασχόληση, δεν είναι δυνατόν να την αποκλείσει, να την αποφύγει. Αυτό το έψκο μόνο μπορεί να το δηλώσει. Βέβαια είναι πολλά τα θέματα που έχουν συζητήσει οι υπουργοί, αλλά για την απασχόληση πρέπει να αφιερώσουν ορισμένοι το χρόνο τους 100% για να βρουν μια λύση και κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο. Να, αυτά. Καλή ήταν νομίζω η ιδέα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ να περιγράψει και τις ελλείψεις, πώς να το πω, αλλά και να κάνει προτάσεις για να ακουστεί καλύτερα. Να εισακουστεί και μάλιστα στην καταλληλότερη στιγμή πριν την Εαρινή Σύνοδο, πριν τη Σύνοδο του Ιουλίου και στη φάση όπου το Δεκέμβριο κάνουμε τον απολογισμό. Έπειτα ακούστηκαν πιο συγκεκριμένες απορίες για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης ή θέσεις πράσινης απασχόλησης. Ε, συζητήσαμε το θέμα με τη Βελγική Προεδρία και συστήσαμε μια ομάδα εργασία στο ΕΜΚΟ για το θέμα που πρέπει να καταλήξει μάλιστα σε μια έκθεση τον επόμενο μήνα για να προετοιμαστούν τα συμπεράσματα του ΕΠΣΚΟ το Δεκέμβριο. Δεν υποκαθιστώ εγώ την Βελγική Προεδρία, αυτό είχε βασιστεί να γνωμοδοτήσει η ΕΜΚΟ το Δεκέμβριο για τις πράσινες θέσεις. Δεν το αγνοούμε λοιπόν ούτε αυτό, αλλά χωρίς να προδικάζω τι θα πούμε στην έκθεση αυτή, θα συζητηθούν μέτρα κατάρτισης, αλλά επίσης και τίθεται ένα θέμα περιγραφής του τι συμβαίνει ως προς την ανάπτυξη οι πράσινες θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να υπάρξουν αν δεν υπάρχουν πράσινα προϊόντα και αν τα πράσινα προϊόντα δεν δημιουργούν πράσινη ανάπτυξη. Αλλά αυτά λοιπόν συνδέονται με όλους τους υπόλοιπους τομείς, όχι μόνο τον μακροχρηματοδοτικό αλλά και τον βιομηχανικής πολιτικής, ανταγωνιστικότητας, έρευνα κλπ. Το συζητάμε, το, το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή και σε λίγο θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Τέλος, για τα κοινωνικά προγράμματα, αν δοθεί όχι προτεραιότητα στο κοινωνική πτυχή μέσω της καλύτερης κατάργησης των μισθωτών αλλά και της στήριξης των εισοδημάτων. Στο έγγραφό μας, μεταξύ των μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης, μαζί με την Κομισιόν λέμε, μιλάμε και για τα μέτρα μερικής ανεργίας και αυτά είναι όλα μέτρα ε, που χορηγούν στον εργαζόμενο μεγαλύτερη ασφάλεια. Υπάρχουν όμως και θέματα ποιότητας της εργασίας, ελκυστικότητας των νέων θέσεων απασχόλησης γιατί και αυτά είναι μία από τις προτεραιότητες της Βελγικής Προεδρίας και τα συζήτησε το ΕΠΣΚΟ. Έγινε μία εξαιρετική διάσκεψη που οργάνωσε η Βελγική Προεδρία. Όλοι λοιπόν συμφώνησαν ότι πρέπει οι νέες θέσεις απασχόλησης να ε, είναι υψηλής ποιότητας. Και άρα επανερχόμαστε έτσι στον τρόπο ενθάρρυνσης της ανάπτυξης δεν πρέπει να ανησυχείτε για αυτά, τα λαμβάνουμε υπόψη. Βέβαια υπάρχουν και τα θέματα των βραχυπρόθεσμων συμβολέων και της ανασφάλειας στην αγορά εργασίας, αλλά και αυτά τα ζητάμε, μην ανησυχείτε. Νομίζω ότι αυτά ήταν όλα και ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκλησή σας και για την ευκαιρία που μου δώσατε εδώ να σας εκθέσω τα σκέψεις μας. Ευχαριστούμε πολύ, ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε για την προσέλευσή σας. Yes, I thought we were missing uh, the rapporteur on the next item, but we're not. Uh, I'll hand straight over for the implementation. Θα περάσουμε αμέσως στην οδηγία για τις ε,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 Θα uh, vous le temps de saluer euh, Θέλω να σας δώσω το λόγο για να αποχαιρετήσω τον κύριο Διευθυντή. Α, σας ευχαριστώ πολύ, λέει πρόεδρος. Λάβε μια σειρά τροπολογιών. Όχι υπερβολικά πολλέ. Υπάρχουν γενικά ευρύτερε δυνατότητε συμβασμών. Δεν θέλω να να αναφερθώ σε κάθε τροπολογία, θα σας αναφέρω μόνο τους αριθμούς. Έχουμε ένα κατάλογο, επιλογή σκέψη α. Νομίζω ότι εκεί είναι δυνατόν να επιτευχθεί σεβασμός μεταξύ των 2, 4 και 5. Για να δω. αναφορά τις πραγματικές θέσεις απασχόλησης. Το 1α. Υπάρχει επίσης νομίζω μια δυνατότητα συμβασμού μεταξύ 8, 9, αυτό το 2. Για το α, α. Εδώ διευκρίνεται ότι ο τομέας των υπηρεσιών α, να λυγεί σήμερα στο 70% θέσεις απασχόλησης και του α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγραφος 1 τώρα. Συμβαστική δυνατότητα μεταξύ της 16, 17 και 18. C'est un peu long, mais il me semble qu'il y a une possibilité 3. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε συμβασμό μεταξύ των 26 και 27.

και 45. Παράγραφος 6. Συμβαστική τροπολογία πάνω κατά την απόψή μου μεταξύ της 50, 51, 52, 53, 54, Αυτά νομίζω. Τα δύσκολα σημεία είναι γνωστά, δεν υπάρχουν εκπλήξεις. το θέμα που αφορά τη γενική εικόνα της ε, οδηγίας για τις υπηρεσίες, δηλαδή τι θα μπορεί να θεωρηθεί ως επιτυχές. Και το δεύτερο, ακαθόδο σημείο, είναι ένα αίτημα που έχουν εκφράσει πολλές πολιτικές ομάδες και πολλοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. της αίτησης ε, οδηγίας πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Έκανα κάποιες προτάσεις για συμβαστικές τροπολογίες. Μπορούμε να επανέλθουμε. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε και να καλύψουμε σε μια θετική απόφαση. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Μου είπαν ότι η τροπολογία 20 έχει κάποιο πρόβλημα σχέση με το κατά πόσο είναι παραδεκτή ή όχι. Φαίνεται ότι βρίσκεται εκτός δικής μας αρμοδιότητας, οπότε δεν είναι παραδεκτή η 20. Αν κύριος Κρίστησαν παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την, την δική του την εργασία και νομίζω ότι πράγματι έκανα μια πολύ καλή δουλειά και νομίζω θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε γενικές γραμμές για την οδηγία αυτή. Θα ήθελα όμως να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ εσφαλμένο εδώ. Επειδή έχουμε εδώ το κατάλογο της ε, ψηφοφορίας με αυτές τις προτάσεις ε, συμβασμού και εγώ παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τον εισηγητή σε αυτά που είπε. Όμως νομίζω θα ήταν σκόπιμο να είχαμε τις προτάσεις αυτές για συμβαστικές τροπολογίες με ένα πιο ξεκάθαρο, πιο σαφή τρόπο. Και μετά για τους μεμονωμένους συμβιβασμούς που ανέφερε ο εισηγητής να πω την άποψη των σοσιαλιστών. Για την εντελογική σκέψη 1 συμφωνούμε στην παράγραφο 1. Ίσως πρέπει να πούμε ότι αυτός ο όρος decent job, αξιοπρεπής εργασία, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη. Αυτό δεν έγινε. Και είπε ότι αν δεν ζητηθεί, δεν γίνεται να προσθέσουμε αυτούς τους όρους. Θεωρώ πάντως ότι αυτό το πρόβλημα θα μπορούσαμε να το λύσουμε και να γίνει κάτι, να βρούμε μια λύση. Μετά έχουμε και την συμβαστική πρόταση για την παράγραφο 3 και εμείς διαφωνούμε εδώ. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τον εισηγητή να εξετάσει όλες τις προτάσεις συμβασμού για την παράγραφο 2 και παράγραφο 3 και ίσως να μπορούσαμε να βρούμε τελικά μια λύση γιατί έχω την εντύπωση ότι κάτι θα βρούμε κατάλληλο στο κείμενο της οδηγίας παρόλο που υπάρχουν κάποια προβλήματα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας έστω και αν υπάρχουν κάποιες μικρές επιφυλάξεις. Τώρα, τούτο λεχθέντος να πω ότι γενικά συμφωνούμε με τις υπόλοιπες προτάσεις της συμβιβαστικέ. Για την παράγραφο 4 τώρα συμφωνούμε για την συμβαστική πρόταση. Βεβαίω, όταν άκουσα την πρόταση του εισηγητή να μην ε, πέταξα τη σκούφια μου αλλά τέλος πάντων όπως έχει αυτή η πρόταση συμβασμού μας βρίσκει σύμφωνος και γενικά χαιρόμαστε που υπάρχει οδηγία σε αυτόν τον τομέα των υπηρεσιών που ρυθμίζονται με αυτόν τον τρόπο. Στην παράγραφο 5 τώρα και στην παράγραφο 6 να πω ότι συμφωνούμε και για τις δύο παραγράφους οι συμβαστικές προτάσεις οπότε αναμένω το αναθεωρημένο κείμενο ώστε να τα βρούμε με τον εισηγητή. Πάντως ε, το ξανά σε γενικές γραμμές συμφωνούμε και θα τα βρούμε με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τούρνεμ, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων κάποια σχόλια. Φαίνεται ότι θα υπάρξει ευρεία συμφωνία στην Επιτροπή μας για τα κύρια ζητήματα. Δύο πράγματα να πω. Καταρχήν να τονίσω αυτό που μόλις υπόθηκε, ότι θα πρέπει και θα εκτιμούσαμε πάρα πολύ στο συμβασμό να υπάρχει ένα συσχετισμό μεταξύ οδηγία των υπηρεσιών και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εργασία ή συμβάσει αυτές των οδηγιών για τις υπηρεσίες. Αυτό νομίζω είναι μια προτεραιότητα και θα μπορούσαμε να βρούμε έτσι μια πιο ισχυρή διατύπωση στο κείμενο. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες γενικού συμφέροντος αυτό είναι ένα τομέα ευαίσθητο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συμφωνήσουμε και να ενισχύσουμε τη διατύπωση, επειδή θα πρέπει να προστατεύσουμε αυτό το είδο υπηρεσιών που είναι γενικού συμφέροντο και έχουν κοινωνικούς σκοπούς ώστε αυτές οι υπηρεσίες να μην υπόκεινται σε νόμους ανταγωνιστικότητας. Θα έπρεπε λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο να το τονίσουμε περισσότερο στην συμβαστική λύση και κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Βλέπω ότι υπάρχουν και άλλες τροπολογίες κατηγορίας ΕΜΚΟ. Οπότε θα πρέπει εδώ να εμβαθύνουμε για το ποιο είναι ο ρόλο τη απασχόληση εδώ. Δεν μιλάω για τη δική σα πρόταση τη συντακτική ή για τι συμβαστικέ προτάσει, αλλά κάποιε τροπολογίε αφορούν αυτό ακριβώ την απασχόληση και ιδιαίτερα τον ρόλο τη Επιτροπή Απασχόληση. Επειδή ακριβώ η ΕΜΚΟ θα ασχοληθεί και με άλλα πράγματα. Και τέλος, μια πληροφορία. Το γνωρίζετε, αλλά στην ΕΜΚΟ, στην Επιτροπή Απασχόλησης, έχει καθυστερήσει η διαδικασία, είμαι μέλος εκεί, οπότε θα υπάρχει εκεί καθυστέρηση. Οπότε είμαστε σε κάποια πρώιμη φάση εδώ. Και συγχαρητήρια για την συμβαστική σας πρόταση και ευχαριστώ για το ανοιχτό δεκτικό σας πνεύμα. Ευχαριστώ, κύριε Στερόσα. Κ. Μπαλτασάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μπαλτασάρ, ναι. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την διαθεσιμότητα που έδειξε και καταγράφω την βούληση για ανέβριση σημείων επαφής και συμβιβασμών για διάφορες, ε, διάφορα σημαντικά στοιχεία της αυτή λοιπόν η πρώτη άθεση μας οδήγησε σε μια συνεργασία και σε μια ανέβρεση έτσι, κοινών σημείων. βεβαίω, εκ μέρου μα υπάρχουν εκ μέρου του ΕΛΚ υπάρχουν και θέσει για τις οποίες δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη δισκαμψία. Ιδιαίτερα για την παράγραφο 1, τροπολογίες 1 με 14, δεν είμαστε έτσι και τόσο σύμφωνοι με την προσέγγιση του εισηγητή. Το ίδιο και στην παράγραφο 3 από το 25 μέχρι το 29 τροπολογίες αυτές τα κριτήρια που επαναλαμβάνουν αυτές οι παράγραφοι δεν τα συμμεριζόμαστε. Και τέλος η παράγραφος 4 που αποτελεί και το κεντρικό ζήτημα προσυζήτηση. Εμείς βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή την ιστορική στιγμή εδώ στο σώμα για το κατά πόσο υπάρχει ανάγκη ή όχι να υπάρχει μια οδηγία που θα ρυθμίζει τις γενικές υπηρεσίες, τις κοινωνικές αλλά και τις γενικότερες φύσεις υπηρεσίες. Έχουμε και τα θέματα της επικορικότητας, οπότε σε αυτό το τομέα θα είναι καλό να αφήσουμε στις χώρες μέλη την δυνατότητα αυτορύθμισης. Αυτά. Κατά τα άλλα, όπου είναι δυνατόν θα συμφωνήσουμε επειδή νομίζω ότι δεν υπάρχουν και έτσι ανυποχώρητα σημεία στις υπόλοιπε παραγράφους, υπάρχει βούληση και εκ μέρους μας, ώστε να καταλήξουμε σε έναν συμβασμό, ώστε να υπάρχει βέβαια αναγνώριση και αποδοχή των ε, αντίστοιχων θέσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο, ε, ο λόγος του εισηγητή στον κύριο Περναμία, ο Σαν Ευχαριστώ πολύ. και εξησεν δεν τελειώσαμε. Γι' αυτό ακριβώς δεν έχουμε κατάλογο ψηφοφορίας. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Έχουμε ακόμα χρόνο μεταξύ μας να ολοκληρώσουμε. Για τις παραγράφους 2 και 3. Γιατί να μην τις ε, διαγράψουμε. Εντάξει, ε, δεν έχω μονομανία, ας το κάνουμε. Τώρα για η αναφορά στην αξιοπρεπή απασχόληση το λέμε στα εκτιμώντας, αλλά θέλετε να παραλαμβάνετε κι αλλού, βεβαίως. Είναι καλό να διευκρινίζουμε και να παραλαμβάνουμε τα πράγματα. Αυτά. Ο συμβασμός λοιπόν δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας να δουλέψουμε. Το λέω αυτό προς όλους τους ομιλητές και ομιλήτριες. Κυρία Τούρινεν, συμφωνώ για αυτό που είπατε προηγουμένω, για να υπάρχει μια διασύνδεση. Να δούμε όμως πώς θα το κάνουμε, ώστε να μην αφαιρέσουμε σαφήνεια από την πρότασή μας. Για τις διευκρινήσεις τώρα για τις κοινωνικές υπηρεσίες, δεν τις διάβασα όλες στο, στην Επιτροπή. Πάντως οι αρχικές προτάσεις συμβασμού τις ανέφεραν και εσείς καταθέσατε προτάσεις ε, επ' αυτού και άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Μπαλτασάρε, σας άκουσα και καταλαβαίνω τι λέτε γιατί εδώ και χρόνια το συζητάμε στο Κοινοβούλιο την έννοια της οδηγίας ε, πλαίσιο για τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος και την επικουρικότητα. Αλλά, αλλά δεν θα πρέπει να το είχαμε πει αυτό από την αρχή ότι θα έπρεπε να κάνουμε διαφορετικά επειδή έχουμε την επικουρικότητα. Πάντω θα πρέπει να δούμε μαζί με εσά και την ομάδα σας τι δυνατότητε υπάρχουν, μέχρι που θα μπορούσατε να πάτε, που δεν θα θέλατε να πάτε καθόλου. Πράγματι, το θέμα της επικουρικότητας αφορά διαφορετικές νοοτροπίες στην Ευρώπη όσον αφορά την έννοια της ε, κοινοφελούς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ε, γενικού συμφέροντος. Θα δούμε λοιπόν σε τι μπορούμε να συμφωνήσουμε σε τι διαφωνούμε, αλλά είμαι πάντως ανοιχτός για οποιαδήποτε συζήτηση. Είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και η βοηθή μου. Είχαμε αρκετές τροπολογίες και ανεξαρτήτως προέλευσης πολιτικής ομάδας νομίζω εύκολα θα βρούμε συμβαστικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. And just to give you some dates... Καλά. Διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη στις Σεπτεμβρίου, στις 23 ε, Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και 8 με 9 Νοεμβρίου στην Επιτροπή θα ζητηθεί και ΕΜΚΟ 30 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν αντιρρήσεις θα ήθελα να περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα, Αμέσω. Διότι οι συντάκτες της μελέτης είναι ήδη παρόντες. Αν έχετε καλέσει κόσμο να ακούσει τη μελέτη και αρχίζουμε νωρίτερα, πέστε το μου να κάνω διάλειμμα. Εγώ προτιμώ να τελειώσουμε νωρίτερα παρά να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Δεν ακούω αντίρρηση. Εγκρίνεται λοιπόν η πρότασή μου. Λοιπόν, η μελέτη λοιπόν για τους αναπήρους και τη συμπερίληψή τους στην αγορά εργασίας ο δόκτωρ Μιχαήλ Κενζήρη και η Βαρβάρα Βαντερουίκη Έχετε αντίτυπα. Έκολ ε, Καντζήρη θα αρχίσει πρώτος λοιπόν. The European Parliament, ladies and gentlemen, thank you very much for giving us uh, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να παρουσιάσουμε αυτή τη στάση για την κινητικότητα και την περίληψη των ανθρώπων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας. Καταρχάς θα ήθελα να κάνω γενικές δηλώσεις το Συμβούλιο της Ευρώπης έθεσε το θέμα των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες και από την κοινωνική χάρτα ήδη από το 1996. Από τότε οι ανάπηροι δεν θεωρούνται πλέον ως ασθενείς ή θύματα, αλλά ως άνθρωποι με ίσα δικαιώματα και πλήρη ρόλο να παίξουν στην κοινωνία. Η στρατηγική της Λισαβόνας και τα κοινωνικά της προγράμματα καθώς και η στρατηγική 2020 έθεσαν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της εξάλληψης της ανέχειας. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί όλο και μεγαλύτερη προσοχή στα κράτη-μέλη στο θέμα της ενδυνάμωσης της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας των αναπήρων ή ανθρώπων με αναπηρίες. Και η μελέτη μας διαπιστώνει ότι ο ρυθμός απασχόλησης των αναπήρων είναι σχεδόν 20% χαμηλότερος από ότι ο ρυθμός απασχόλησης των μη αναπήρων, των αρτιμελών. Και το μορφωτικό τους επίπεδο των αναπήρων είναι επίσης χαμηλότερο από ότι εκείνο των αρτιμελών. Εδώ οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη ως προς τους αναπήρους είναι η χαμηλή τους απασχολησιμότητα, η υψηλή εξάρτηση από επιχορηγήσεις, περισσότερες δημόσιες δαπάνες και μεγαλύτερος κίνδυνος να βρεθούν κάτω από το όριο της ανεχίας. Η διανοητική αναπηρία ή ασθένεια είναι ο κυριότερος λόγος που προβάλλεται για την μη απασχόλησή τους. Και ακόμη και αν τα διανοητικά αυτά προβλήματα είναι μέτρια όπως ε, κατάθλιψη. Όλες σχεδόν οι αιτήσει για αποζημιώσεις αναπηρίας σχετίζονται με τέτοια διανοητικά προβλήματα. Μεγάλος αριθμός νέων κάτω των 35 ετών που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας έχουν σημειωθεί σε όλες τις χώρες μέλη. Και αυτό είναι πολύ ενισχυτικό. Διότι παραδοσιακά κάποιος που δέχεται επίδομα αναπηρίας ήταν αρσενικό άτομο μεγαλύτερης ηλικίας με χειρονακτική εργασία και έπαιρνε αυτά τα επιδόματα ως πρόγραμμα πρώιμης συνταξιοδότησης ας πούμε. Αλλά η τάση αυτή αλλάζει τώρα και είναι όλο και περισσότεροι οι νέοι. Και αυτό είπαμε ότι είναι ανησυχητικό διότι τα επιδόματα αναπηρίας θεωρούνται ακόμη στην Ένωση ως ε, ως συντάξει σε φόρο Δηλαδή ένας νέος που αρχίζει να παίρνει ένα τέτοιο πρόγραμμα επιδόματος μάλλον θα αποκλειστεί καθόλου του τη ζωή από την αγορά εργασίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις η δυνατότητά τους για εργασία τμηματικά, μερικά μόνο μειώνεται στην πραγματικότητα. Στο πίνακα 6 βλέπετε ότι οι ανάπηροι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να βρεθούν κάτω από το όριο της ανέχειας εφόσον μάλιστα δεν απασχολούνται. Στον πίνακα 2 στον διεφαίνεται το ποσοστό των νέων επιδομάτων που χορηγούνται λόγω κακής διανοητικής υγείας. Κάτι άλλο, η κινητικότητα των αναπήρων. Η κινητικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσει η εργατική δύναμη της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις ε, συνεχώς αλλάζουσες συνθήκες της αγοράς. Παραδοσιακή φραγμή όπως νομική ή διοικητική είναι πολύ βαρύτερη και αρνητικότερη για τους αναπήρους. Η μελέτη μας ταύτισε πολλές αναπηρίες που δίνουν δικαίωμα σε επιχορηγήμουσης. Αυτό θέτει ορισμένα προβλήματα όταν συζητούμε το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας. Γιατί όσοι έχουν κάποια αναπηρία δεν τους εφαρμόζονται οι ίδιοι ορισμοί και τα κριτήρια σε ολόκληρη την Ένωση. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μου που θα σας περιγράψει τα μέτρα που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανθρώπων με αναπηρίες. Τι είναι συνάδελφό μου. Καλησπέρα σας. Γενικά υπάρχουν δύο είδη μέτρων για τα άτομα με αναπηρία. Αφενός παθητικά μέτρα που αφορούν επιδόματα και αφετέρου ενεργικά μέτρα με ενεργές δηλαδή πολιτικές απασχόλησης. Στα δεύτερα έχουμε κάνει μια διάκριση σε τρία είδη κατηγοριών ανάλογα με τους ανάπηρους. Η πρώτη κατηγορία είναι ενημέρωση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ψυχολογική καθοδήγηση. Η δεύτερη κατηγορία είναι κατάρτιση και επιμόρφωση, εκπαίδευση κλπ. Και η τρίτη κατηγορία αφορά την ανέβρεση εργασίας. Προστατευόμενη μορφή εργασίας όπως έχουμε σε χώρες Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία κλπ. Δύο είδη μέτρων απασχόλησης επίσης αναφέρονται. Αφενός έχουμε συγκεκριμένα μέτρα, δηλαδή αυτά που στοχεύουν σε ανάπερους ε, ανθρώπους, όπως συστήματα ποσοστώσεων που υπάρχουν στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μόνο η Δανία και η Φιλανδία δεν έχουν συστήματα ποσοστώσεων για τους ανθρώπους με αναπηρία. Στον πίνακα εδώ στο 13 και στο 14 θα βρείτε κάποια παραδείγματα των συστημάτων με ποσόστοση και σε κάποιες χώρες αυτό συνδυάζεται με κάποιες κυρώσεις, σε άλλες όχι. Ένα άλλο είδος μέτρων απασχόλησης αφορά κάποια γενικότερα μέτρα όπως πολιτικές κατά της διάκρισης, όπως και μέτρα προσβασιμότητας, δηλαδή προσαρμογή στον χώρο της εργασίας, κάτι το οποίο αφορά περισσότερο την φυσική προσαρμογή, προσαρμογή στις συνθήκες εργασίας όπως ευελιξία και προσβασιμότητα στην πληροφόρηση. Ένα τρίτο είδος γενικών μέτρων είναι το flexicurity. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό επειδή βοηθάει στο να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ των ενεργητικών και υποθετικών μέτρων και να βρούμε επίσης ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και απασχόλησης. Όμως όλα αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς μια θεσμική μεταρρύθμιση όπως αυτή που έγινε στην Δανία. Το πρόγραμμα για την αναπηρία στην Δανία μεταρρυθμίστηκε το 2003 και δόθηκε έμφαση όχι πια στο τι μπορεί να κάνει ένα άτομο και όχι στο τι δεν μπορεί να κάνει. Οπότε δηλαδή φύγαμε από την νοοτροπία και την κουλτούρα της αναπηρίας και πήγαμε στην ε, νοοτροπία και στην κουλτούρα των δεξιοτήτων. Όσον αφορά τώρα τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο αυτών των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν, είναι δύσκολο να αποτιμηθεί επειδή υπάρχει έλλειψη στοιχείων σχετικά με τα μέτρα αυτά. Οπότε η γνώση μας είναι αρκετά περιορισμένη. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν διάφοροι φραγμοί όσον αφορά την σωστή εφαρμογή των μέτρων όπως περιορισμένοι πόροι, έλλειψη διαθέσιμων πληροφοριών, έλλειψη οικονομικών στοιχείων, έλλειψη στοιχείων από άτομα με ειδικέ αναπηρίες, ε, ε, έλλειψη στοιχείων από τους εργοδότες κλπ. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οριστικά όσον αφορά και τους φραγμούς και είναι δύσκολο να κάνουμε μια αποτίμηση εκεί. Βεβαίως ε, είναι δύσκολο να πούμε κάτι όταν έχουμε αρκετά τεκμηριωμένα στοιχεία στη διάθεσή μας. Όμως μπορούμε να πούμε ότι τα συστήματα με ποσοστώσεις βοηθούν, όμως βοηθούν αυτούς που ήδη έχουν δυνατότητα ανέβρεσης θέσης εργασίας. Ξέρουμε επίσης ότι ένα συνεκτικός συνδυασμό μέτρων θεωρείται να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, όπως ένας συνδυασμό μέτρων και νομοθεσιών κατά των διακρίσεων με απαιτήσει για τους εργοδότες να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές στον χώρο της εργασίας. Το flexicurity αποτελεί επίση άλλη μια πολύ σημαντική πτυχή και θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την περίληψη, ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίε στην, ε, στην αγορά εργασία. και ο συνάδελφό μου θα, και πάλι θα σα αναφέρει κάποιε συστάσει. Προσπαθήσαμε να ε, διατυπώσουμε 7 ε, συστάσεις το τρίτο θέμα της παρουσίας μας, καταρχήν όσον αφορά τον τίτλο κινητικότητα και ένα ατόμων αναπηρία στην αγορά εργασία. Το θέμα της εφαρμογή τη νομοθεσία των μη διακρίσεων μέσα στην νομοθεσία τη κοινοτητα ήταν ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι γι' αυτό πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ε, διασφαλίσει η αρχή αυτή να εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να τονίσει στην επόμενη του έκθεση για τα θέματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες ότι πολιτικές μεταρρυθμίσεις συστημάτων επιδοτήσεων στα κράτη-μέλη θα πρέπει να βασίζονται στη δυνατότητα εργασίας και όχι στην αδυναμία εργασίας ατόμων με αναπηρίες. Είναι βέβαια σημαντικό και απαραίτητο να προστατεύσουμε εκείνους που είναι ασθενείς ή τραυματίες. Από την άλλη μεριά, τα συστήματα ωφέλης είναι να ε, υποστηρίζουν εκείνους που μπορούν να εργαστούν για να παραμείνουν στην αγορά απασχόλησης. Ε, αντί δηλαδή να συνεχίσουμε με το status quo, θα πρέπει να προωθήσουμε μία ε, πολιτική ένταξης. Εκτός αυτού, πιο ευρύς πολιτικές θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να αποφευθεί η παγίδα των επιδοτήσεων αναπηρίας, παραδείγματο χάρη, με την ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων στον ιατροφαρμακευτικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τους νέους το πρόβλημα της πνευματικής υγείας των νέων είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για το μέλλον, γιατί πολλοί από αυτούς ε, παραμένουν παγιδευμένοι, αν θέλετε, ε, στον τομέα των επιδοτήσεων αναπηρίας και δεν, μόνο το 3% επανεντάσσονται στο χώρο απασχόλησης. Εμείς λοιπόν αναλύουμε τις μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά να παραμείνουν εν ενεργεία. Μια κοινωνική, ένας κοινωνικός συνασπισμός θα μπορούσε να βοηθήσει και να καταστήσει την εργασία πιο προσφυλή προς την υγεία. Η προσέγγιση της ευελιξίας με ασφάλεια, security, θα πρέπει να έχει θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση ατόμων με αναπηρίες ιδίως ευέλικτα προγράμματα εργασίας, μέτρα ενεργοποίησης, ταυτόχρονα με συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που εξασφαλίζουν αποδεκτά επίπεδα διαβίωσης, νομίζω ότι είναι κάτι που το χρειαζόμαστε. Μια που δεν έχουμε πολλά εμπειρικά στοιχεία, δεν μπορούμε να πούμε κατά πόσον το ένα μέτρο είναι το σωστό και το άλλο λιγότερο σωστό όσον αφορά την ένταξη των ατόμων αυτών με τις αναπηρίες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να είναι υπέρ ενός προτύπου flexicurity, δηλαδή ένα μέγεθος για όλους, Τον αντίον θα πρέπει να προωθεί την βασική ιδέα της ευελιξίας με ασφάλεια της flexicurity. Επίσης, όπως είπα ήδη, από τη μελέτη μας είδαμε ότι δεν έχουμε αρκετά εμπειρικά στοιχεία όσον αφορά την ε, επιτήρηση και αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης ατόμων με ειδικέ ανάγκες. Η στολική στοιχείων και η πρόσβαση στη γνώση για τις βέλτιστες πρακτικές θα βοηθήσουν να ερευνηθούν οι καλύτερες μεθόδους, συγγνώμη, για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την συλλογή και παρουσίαση των στοιχείων αυτών. Ιδίω έχω κατά νου μια εναρμοσμένη ε, μορφή συλλογής στοιχείων. οι διάφορες πρωτοβουλίες πολιτικές που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα μπορούν να συνεργαστούν εναρμονισμένα μόνο εισαγάγοντας ένα υψηλό επίπεδο συνέπειας. Η κλίδα για να επιτευχθεί αυτό είναι βελτιωμένη επικοινωνία. Όχι μόνο μεταξύ διαφόρων κοινοτικών οργάνων και σωμάτων, αλλά και στο εσωτερικό τους. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βοηθήσει να υπάρξει καλύτερος συσχετισμός μεταξύ των εθνικών πολιτικών απασχόλησης και των εθνικών πολιτικών για την κοινωνική ένταξη. Η τελευταία σύσταση πολιτικής που έχω να κάνω αφορά το επόμενο πρόγραμμα δράσης για την αναπηρία χρησιμοποιώντας ισχύουσες μεθόδους συντονισμού στον τομέα της απασχόλησης, πράγμα που θα μπορούσε να βοηθήσει ούτως ώστε τα θέματα της ε, αναπηρίας να συζητιούνται πιο συχνά από τους νομοθέτες σε εθνικό και σε κοινωτικό επίπεδο. Ο στόχος της πρόθεσης ανεξάρτητης κατοικίας για τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να είναι θεματική προτεραιότητα στο επόμενο πρόγραμμα δράσης για τους αναπήρους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Αυτά έχουμε να πούμε εμείς και περιμένουμε να ακούσουμε τις ε, απόψεις μεγάλων ενδιαφέρον. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ χρήσιμο όλα αυτά και σας ευχαριστώ για το έργο που επιτελέσετε. Πριν δώσω το λόγο σε οποιοδήποτε άλλο, έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις που θα ήθελα να μου επιτρέψετε να υποβάλω και κάποια σχόλια. αναφερθήκατε στη δυσκολία που υπάρχει γιατί κάθε κράτος μόνος έχει διαφορετικό ορισμό της αναπηρίας. Και εγώ πάντα θεωρούσα αυτό το πρόβλημα τεράστιο. Και όπως ε, ξέρετε καταφέραμε στην ε, Euro Convention να καταλήξουμε σε έναν ορισμό για την αναπηρία. Αυτού του τύπου τον, ε, την προσέγγιση θέλετε να δείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ορισμό για την αναπηρία βασιζόμενο στον ορισμό της Convention. Επίσης, αναφερθήκατε στο θέμα της ε, δυνατότητας πρόσβασης. Έχουμε βέβαια εμεί αυτή την οδηγία που προβλέπει γενικά δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό χώρα απασχόληση. Μπορείτε να μας αναπτύξετε πώς πιστεύετε ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την οδηγία αυτή. Ξέρω ότι η Κομισιόν έχει εισακάγει κάποιε διαδικασίε επί παραβάση για κάποια κρατημέλη σχετικά εδώ, αλλά πιστεύετε ότι εξακολουθεί πραγματικά να μην έφταναν σωστά στα διάφορα κρατημέλη. Πολλοί το κάνουν, αλλά μόνο από εδώ και από εκεί δεν υπάρχει τίποτα έτσι ενιαίο. Ποια είναι τα προβλήματα και πώ πιστεύετε ότι πρέπει να επιληθούν. Τούτου λεχθόντος για το θέμα τη πρόσβαση. Από όσο βλέπω στην εκθεσή σας, δεν ασχοληθήκατε με το θέμα της ε, δυνατότητας πρόσβασης στον τόπο απασχόλησης. Γιατί βέβαια έχουμε και την οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων που θα πρέπει να επιτρέψει τη δυνατότητα πρόσβασης στα κτίρια, στα μέσα μεταφοράς και σε διάφορες δομές και πόσο σημαντικό θεωρείτε εσείς αυτό το τομέα. Δηλαδή να μπορούν όλοι να έχουν δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τον τόπο απασχόλησή του. Και όχι μόνο το θέμα τη πρόσβαση μια φορά μετά που θα φτάσουν. Τέλο, στο τέλο τη παρουσίαση σα αναφερθήκατε στο θέμα τη ανεξάρτητη διαβίωση και κατοικία. Έχετε κάποια μελέτη πώ αυτό βοηθάει του αναπήρους για να είναι πιο ικανοί να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας αργότερα. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί που ζουν πραγματικά ανεξάρτητα και όχι σε ιδρύματα μπορούν πολύ πιο εύκολα να εργαστούν γιατί αισθάνονται πιο ικανή προς εργασία. Άλλο αυτό. Και ενδιαφέροντα στοιχεία μας δώσατε για τα άτομα με πνευματικές αναπηρίες. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ειδικό πρόβλημα. γιατί πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το θέμα της ε, πνευματικής αναπηρίας είναι κάτι που θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε. Και όπως είπα θα πρέπει να το εξετάσουμε έγκαιρα. Μπορείτε να αναπτύξετε και αυτό το θέμα. Γιατί ξέρω ότι όταν κάποιοι έχουν αρχίσει να εργάζονται και εξακολουθούν όμως να διώκονται από τα προβλήματα της πνευματικής τους αναπηρίας, έχουν περισσότερο στρες στην θέση απασχόλησης. Και επίση μπορώ να σα υποστηρίξω με αυτά που είπατε για την flexicurity, για την ασφάλεια με ευελιξία. Πρέπει πραγματικά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ευελιξία στην εργασία του, ούτω ώστε να μπορούν τα άτομα αυτά κάποια φορά να εργάζονται μερική απασχόληση, να φύγουν, να ξανάρθουν. Και βέβαια, όταν αυτό ορισμένοι είναι περιορισμένοι στα επιδόματα. λοιπόν δεν μπορούσαμε να το μέχρι στιγμής να το προβάλλουμε στην οθόνη. Τώρα μπορούμε, αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε. Και αυτό που μου είπατε εσείς είναι ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ε, αυτοί οι άνθρωποι να ενθαρρυνθούν να εργαστούν παίρνοντα τα επιδόματά τους ακόμα και όταν εργάζονται. Να τους ενθαρρύνουμε κατά τον τρόπο να εργαστούν. Ιδίω αν κάποιος ε, γίνει ανάπηρος λόγω μια ε, ασθένεια ή δυστυχήματος. και τα άτομα αυτά δεν αισθάνονται ικανοί ή δεν αισθάνονται ότι θα μπορούσαν πραγματικά να επανέλθουν στον τόπο εργασίας τους. Έχουν αντίποση, δηλαδή όταν έχουν πάθει ένα δυστύχημα στην εργασία τους, έχει κλείσει η πόρτα, δεν αισθανονται οτι θα μπορουσαν πραγματικα να ερθουν στον τοπο εργασιας τους εχουν εντυπωση δηλαδη οταν εχουν παθει ενα δυστυχημα στην εργασια τους εχει κλεισει η πορτα δεν μπορουν πια να ξαναεργαστούν. Αυτά, στα τα δικά μου σχόλια, ο κύριος Κώστα νομίζω ότι είναι επόμενος. Παρακαλώ. Thank you. Adam Köszönöm a Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συντάκτες αυτής της έκθεσης που αποτελεί μια, μια θαυμάσια κίνηση, ένα θαυμάσιο σημείο κίνησης. Εγώ διάβασα την έκθεση αυτή και σχημάτισα την εντύπωση την πρώτη εντύπωση ότι τα συμπεράσματά σας όσον αφορά τα συστήματα ποσοστώσεων ότι είναι προσωρινά. Νομίζω ότι έχετε μάλλον κάποιες επιφυλάξει, κάποια έτσι αρνητική στάση σχέση με τα προγράμματα που περιλαμβάνουν ποσοστώσεις. Οπότε ποια θα ήταν η λύση σε αυτό το σημείο προσωπικά εγώ είμαι υπέρ αυτών των προγραμμάτων με ποσοστώσεις γιατί έχουμε κάποια άτομα ε, στο εσωτερικό αυτών των ομάδων ατόμων με αναπηρία τα οποία νομίζω δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στην εργασία χωρίς ε, αυτή ακριβώς τη βοήθεια. Και το δεύτερο μου ερώτημα είναι το ότι ενδεχομένως δεν έχει δοθεί αρκετή σημασία στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο ομάδες στο εσωτερικό αυτό που της ομάδας αυτής που ονομάζουμε άτομα με αναπηρία. Εγώ έχω πτυχίο, έχω επαγγελματική εμπειρία και μπορώ να ανταγωνιστώ αυτούς που έχουν πλήρες δεξιότητες στον τομέα της εργασίας. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν κάποια μορφή αναπηρίας και οι οποίοι δεν είναι σε θέση να λάβουν κάποια εκπαίδευση ή να αποκτήσουν δεξιότητες και αυτή είναι η πλειοψηφία. Νομίζω λοιπόν ότι όπως και οι συντάκτες το σύμφωνο αναπηρίας είναι κάτι πολύ σημαντικό θα πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής 2020 και πιστεύω ότι δεν έχει δοθεί αρκετή προσοχή στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αναφερθήκατε στην ε, συνθήκη του ΟΗΕ, πολύ ωραία, όμως είναι εξίσου σημαντική, αν όχι σημαντικότερη, και χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων της συνθήκης Λισαβόνας. Εγώ δεν είδα να γίνεται κάποια περιγραφή μιας μεθόδου ή μιας ε, μεθοδολογίας για την αύξηση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία. Γνωρίζω ότι αυτά τα θέματα σχετίζονται με νομοθεσία που αφορά τον ανταγωνισμό, τις δημόσιες προμήθειες, τις, τις δημόσιες, διαγωνισμούς, συγγνώμη, πολιτική δημοσίων διαγωνισμών, δημόσια διαγωνισμοί που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν άτομα με αναπηρία. Δεν ξέρω, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο ως, ως ιδέα. Πάντως συμφωνώ με την Πρόεδρο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ορισμού. Δηλαδή υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό των χωρών μελών και συμφωνώ επίσης με την Προεδρεύουσα ότι η σύμβαση του ΟΗΕ είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να βρούμε ορισμό στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. κυρία Μέσναρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ε, τον ε, ε, κύριο που παρουσίασε την ε, μελέτη. της στην στην γιατί έζησε ένα χάος στο σταθμό στις Βρυξέλλες ε, φτάνοντας εδώ. Συμβαίνει και αυτό φαίνεται θα πρέπει να αναφερόμαστε πραγματικά όχι στην αναπηρία, στο τι δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο άνθρωπο αυτό, αλλά σε αυτό που μπορεί να κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το μέλλον τη αγορά απασχόληση. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε, από τη μια μεριά θέλουμε οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν περισσότερο από ό,τι μέχρι στιγμή και έτσι στο μέλλον θα έχουμε, μια που ο πληθυσμό τη Ευρώπη, ένα μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων με αναπηρίες γιατί σήμερα λόγω της ε, ιατρικής πρόοδου επιζούν περισσότερα παιδιά με αναπηρίες ακόμη και με σοβαρές αναπηρίες. Ένα αυτό το άλλο είναι που το αναφέρετε εξής, ότι ορισμένοι έχουν δυστυχήματα στον ε, χώρο εργασίας ή και ψυχολογικά με το burnout ε, βγαίνουν από τον χώρο εργασίας και θα πρέπει κάπως να φροντίσουμε να ξαναμπούν. Δηλαδή όλα τα άτομα αυτά με αναπηρίες ή ε, με κάποιες προσωρινές, ε, κάποια προσωρινά προβλήματα ε, παραμένουν σε μια παράλληλη αγορά εργασίας, πράγμα που δεν θα είναι καθόλου καλό. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε το περισσότερο να μπορούν να συμμετέχουν στην πρώτη αγορά εργασίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές μορφές απασχολής στην πρώτη αγορά εργασίας. Και νομίζω ότι αυτή η έκθεση πραγματικά ε, ενδείχνεται πάρα πολύ για να σκεφτούμε τα πράγματα αυτά. Και το δεύτερο για την κινητικότητα. Εγώ είμαι και στην Επιτροπή Μεταφορών, όπου ακριβώς συζητάμε αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα των ταξιδιωτών στις μεταφορές με πούλμαν και εκεί παίζει σημαντικό ρόλο το θέμα των αναπηριών. Ε, πράγμα που δεν μπορούμε να λάβουμε τόσο πολύ υπόψη ίσως τα λεωφορεία τα αστικά, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει πραγματικά να είναι κάτι που να μας απασχολεί όσο πάει και περισσότερο. Ευχαριστώ όλοι Tak Ευχαριστώ. και ευχαριστώ πολύ για αυτές τις δύο παρουσιάσεις, για αυτό το σημαντικό ζήτημα. Νομίζω ότι είναι αναφυσβήτητο ότι σε περίοδους ε, κρίσεως όπως αυτή που διανύουμε οι πιο αδύναμοι υποφέρουν και γι' αυτό ακριβώ το λόγο θα πρέπει να κάνουμε στατιστικές για την περίοδο 2008-2009-2010 και θα δούμε εκεί ενδεχομένως ότι οι άνθρωποι με αναπηρία έχασαν, είχαν τις μεγαλύτερες απώλειες ήταν οι μεγάλοι χαμένοι από την κρίση αυτή τα τελευταία χρόνια. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ένα ενιαίο μοντέλο ή μια ενιαία λύση στις διάφορες χώρες μέλη. Επειδή υπάρχουν διάφορες καταστάσεις και διαφορετική βαθμή ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, θεωρώ ότι εξάλλου υπογραμμίζουμε υπερβολικά το θέμα του flexicurity. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ευελιξία, ακριβώ για να επιτρέπουμε την επανένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασία. Όμω αυτό που ονομάζουμε ενεργό πολιτική τη ε, αγορά εργασία είναι πιο σημαντικό δεν έχουμε να κάνουμε λοιπόν μόνο με το flexicurity. Θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ανάγκε τη αγορά εργασία και θα πρέπει να δούμε ακριβώ και τι δεξιότητε και τα ατού, τα πλεονεκτήματα των ατόμων με αναπηρία, ώστε να βρούμε ένα κοινό σημείο, ένα σημείο επαφή. Εδώ ακριβώ θα πρέπει να υπάρχει το flexicurity. Αυτό ακριβώ είναι η καλή πολιτική στον τομέα τη αγορά εργασία. Εγώ γνωρίζω μια κατάσταση που επικρατεί στην ε, Δανία δηλαδή και γνωρίζω πολύ καλά ότι επί παραδείγματι κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε μπορεί κανείς να είναι άνεργος και να έχει δικαίωμα για διάφορα επιδόματα. Υπάρχουν ταυτόχρονα όμως συγκεκριμένα μέτρα τα οποία επιτρέπουν στο άτομο με αναπηρία να μην εργάζεται καθημερινά. Ωραία το flexicurity, πολύ ωραία, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ενεργό στην αγορά εργασίας, ώστε να επιτρέψουμε

είναι προφανές ότι χρειάζονται, ότι πρέπει και οι άνθρωποι με αναπηρίες να μπορέσουν να μπουν στην αγορά εργασίας και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται κατάρτιση. Αυτό είναι ένα από τους κύριους λόγους χρήσης των κοινωνικών ταμείων. Και έχω ακούσει πολλούς ανάπηρους να μου λένε ότι δεν χρησιμοποιούνται όσο θα μπορούσαν. Γιατί, διότι πολλές φορές τα προγράμματα που υποβάλλουν οργανώσεις που τους εκπροσωπούν δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικά. ανταγωνιστικά. Και στις προτάσεις τους, στα σχέδιά τους, στα προγράμματά τους αντιμετωπίζεται μόνο το πρόβλημα του πρόσθετου κόστους που θα επιφέρει η χρήση ανθρώπου με αναπηρίες ή ανθρώπων με αναπηρία και θα χρειαστεί μεγαλύτερη, περισσότερη κατάρτιση ειδική χώρη καμιά φορά και προβλήματα στις μεταφορές τους, τη μεταφορά τους. Τα κοινωνικά ταμεία βέβαια ε, αυτό ακριβώς στοχεύουν. Πώς θα διευκολύνουν την πρόσβαση ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Η κυρία Χανίλσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα Ολλανδικά, αν δεν απατώμε. Πριν εκλεγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ήμουν διευθύντρια της ε, Ολλανδικής Υπηρεσίας Ίσης Μεταχείρισης και πολλές φορές μου έγραφαν άνθρωποι με αναπηρίες ότι τους έχουν αρνηθεί θέσεις Μόλις ο εργοδότης έβλεπε ότι ο υποψήφιος είναι ανάπηρος, αρνούνταν. Έλεγε, α, δεν μπορεί να δουλεύει κανείς σε παιδικό σταθμό ως ανάπηρος, ας πούμε. Και όποτε είχα αναλάβει μια υπόθεση, τόνιζα ότι υπάρχουν μέτρα ίσης μεταχείρισης και ότι πρέπει ο εργοδότης να το ξανασκεφτεί. Πρέπει λοιπόν αυτό να κάνουμε, να τονίζουμε την ε, ευθύνη που έχει ο εργοδότης. Η ε, νομοθεσία ίσης μεταχείρισης πρέπει να εφαρμόζεται. Και όποτε απαιτείται να τους προσάγουμε στο δικαστήριο. Πρέπει να συνεχίζουμε να τονίζουμε ότι καλό είναι, καλό είναι να προειδοποιούμε τον εργοδότη ότι η διαφοροποίηση στον τόπο εργασίας είναι κάτι θετικό. Πρέπει λοιπόν αυτό να το ενθαρρύνουμε ώστε να εφαρμόζεται σωστότερα και καλύτερα η νομοθεσία που υπάρχει για ίση μεταχείριση. Αν έχει κανείς μια αναπηρία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όλα μπορεί να τα κάνει σχεδόν. Ευχαριστώ. Με ορισμένε προσαρμογέ. Δεν νομίζω ότι έχει ζητήσει κανεί άλλο το λόγο. Οπότε επιστρέφουμε στους συντάκτες της μελέτης τον Μιχαήλ και τη Βαρβάρα. Και Τζία και Βαντερβέκ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά είπατε. Ας αρχίσω με την κυρία Λίντσε. Περιορισμών. Το ψήφισμά σας, κυρία Λίνεν, το 2006, στο ψήφισμά σας ήδη ζητούσατε έναν κοινό ευρωπαϊκό ορισμό πριν από τέσσερα χρόνια. Και συμφωνούμε απόλυτα. Ίσως πρόκειται για θέμα έλλειψης σύγκλησης. Η ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων με αναπηρίες είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Πρέπει να μπορούν να μετακινηθούν από μια χώρα στην άλλη. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει ακόμη κάτι τέτοιο επειδή δεν τους εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια και οι ίδιοι ορισμοί σε ολόκληρη την Ένωση. Συμφωνούμε λοιπόν επ' αυτού. Και έχετε δίκιο, η σύμβαση του ΟΗΕ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κατάλληλο βήμα. Απ' τη μία πρόκειται για ανθρώπινο πρόβλημα, δηλαδή οι άνθρωποι με αναπηρίες έχουν και αυτοί δικαιώματα και ευκαιρίες και απ' την άλλη οικονομικά θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ρυθμό απασχόλησης με τη χρησιμοποίησή τους. Η συμπερίληψη λοιπόν και των αναπήρων στην αγορά εργασίας είναι θέμα ζωτικό διότι μειώνεται έτσι και ο κίνδυνος να πέσει κανείς κάτω από το όριο της ανέχειας. Ένα άλλο τώρα εδώ ε, ο συνδυασμός ναι, εμείς δεν λέμε ότι... Εμείς δεν λέμε ότι λέγω χρειάζονται ποσοστώσεις, αλλά αντίθετα θεωρούμε ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας Υπάρχουν πολύ λίγες μάλλον θέσεις εργασίας για ανθρώπους με μικρή κατάρτιση. Εμείς θα θέλαμε να υπάρξει ένας συνδυασμός μέτρων ενεργοποίησης που είπανε σωστής κοινωνικής ασφάλισης, λογικού βιωτικού επίπεδου και ευελίκτων προγραμμάτων απασχόλησης. Όσοι έχουν κάποια αναπηρία και θέλουν να συμμετάσχουν στην αγορά εργασίας, δεν πρέπει να την χάνουν κιμβινέ. Όταν εργάζονται μερικό και όχι μεταχείρισης ή να κινδυνεύουν όταν εργάζονται μερικός και όχι πλήρως ας πούμε. Τι άλλο, αν ναι. Η αναθεώρηση της τάσης μας. Ίσα δικαιώματα σημαίνουν ίσες ευκαιρίες, το είπα και πριν. Και φυσικά πρέπει να ξαναδούμε, να ξανασκεφτούμε το παλαιότερο πρότυπο που ίσχυε. Γιατί σας είχα πει ότι χαρακτηριστικά αυτός που έπαιρνε επίδομα αναπηρίας ήταν άντρας μεγαλύτερης ηλικίας σε κάποια χειρονακτική θέση. Αλλά αυτό δεν ισχύει πια αλλάζουν τα πράγματα. Είναι περισσότεροι νέοι με αναπηρίες. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε περισσότερο τη δυνατότητα απασχόλησης και όχι την αδυναμία απασχόλησης. Όπως κάνει παραδείγματος χάρη η δενημαρκία Και για μας είναι ίσως η βέλτιστη πρακτική που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άλλο τα στοιχεία για την κρίση πρέπει να δείξουμε, επιδείξουμε υπομονή γιατί τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί με βάση την κρίση και τις επιπτώσεις της και στην απασχόληση των αναπήρων από το 8 μέχρι το 11. Θα έρθουν όμως και θα τα δούμε και αυτά. Τώρα για την πρόσβαση και τις ποσοστώσεις θα ήθελα να σας μιλήσει η Βαρβάρα. Ναι, για την πρόσβαση και την προσβασιμότητα. Πολύ και κυρία δεν χρειαζόμαστε μόνο Αλλαγέ στο χώρο εργασία, αλλά βέβαια θα πρέπει να ζητήσουμε και αλλαγέ στην πρόσβαση στο χώρο εργασία, όπως αλλαγές στα μέσα μεταφοράς. Νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε και με άλλε μορφέ εργασία, όπως η τηλεργασία ή η εργασία εξ αποστάσεω. όπου θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος συνδυασμού μέτρων προσαρμογής για τα άτομα με αναπηρίες, για την ε, μεταφορά, αλλά και για την εργασία όταν γίνεται αυτή από, τον, από το σπίτι τους. Αυτά έχω να πω εγώ. Ναι, νομίζω ότι καλύψατε περισσότερα από τα ερωτήματα τα οποία ανέκυψαν, εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που νομίζει ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημά του. Να πω πάντως ότι κάνετε μια πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μελέτη και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στην πρόεδρο μας την κυρία Μπερές. Euh, euh, Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ την αντιπρόεδρο που μου αντικατέστησε. Ήμουνα στην Κόζακ. Θα περάσω, θα περάσω στο σημείο 8 της ημερήσιας. 7. Λέει η ημερήσια όπου η κυρία Καρυματελή θα μας παρουσιάσει το κείμενο το οποίο αφορά την απελευθέρωση του νομικού των κλάδων, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Ε, κύριε Σεχήτρη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν να σας παρουσιάσω τις κύριες γραμμές της γνωμοδότησής μου σε σχέση με την πράσινη βίβλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ω τίτλο Απελευθέρωση του νομικού του κλάδου πολιτισμού και τη δημιουργικότητα, θα ήθελα εδώ να σα εκφράσω την αγανάκτησή μου για την απέλαση που είχαμε το Σαββατοκύριακο 30 νέων φοιτητών που είχαν καταλάβει ένα κτίριο εδώ και αρκετό καιρό κτίριο το οποίο ήταν κενό εδώ και 40 χρόνια στην πλατεία Βόση στο Παρίσι. Αυτοί δεν είχαν που να κοιμηθούν και εγώ δεν μπορώ να σταθώ δίπλα τους σήμερα. Θα ήθελα όμως να εκφράσω όλη την αλληλεγγύη μας ενώπιον αυτών το, αυτής της κατάστασης της κρίσης τα πρώτα θύματα ήταν αυτοί. Ζητάω από τον αρμόδιο Γάλλο Υπουργό Κατοικίας να τους βρει κατάλημα και νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να να εκφράσουμε αλληλεγγύη και να μην ε, παραγνωρίζουμε παραβλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στους δρόμους μας. Τώρα για την ουσία της γνωμοδότησής μου. Νομίζω ότι η βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελούν μία αναφορά, όπως λέει, αποτελούν μάλλον ένα στοιχείο, όπως λέει η πράσινη βίβλος της Κομισιόν, ένα στοιχείο ανταγωνιστικότητας, ανταγωνιστικότητας που θα πρέπει να τονιστεί εν ώψη της στρατηγικής 2020. Νομίζω λοιπόν ότι ο τομέας του πολιτισμού και της δημιουργικότητας είναι και ένας τομέας όπου ισχύει και βασιλεύει μια ποικιλομορφία μορφών εργασίας και καταστάσεων με μεγάλες κοινωνικές ανισότητες για πάρα πολλούς εργαζόμενους. Γι' αυτό ακριβώς επιμείναμε για την ανάγκη μείωσης των ανισοτήτων στον τομέα αυτό. Όχι μόνο των οικονομικών, αλλά και της πρόσβασης στα, στο δίκαιο εργασίας και στην κοινωνική πρόνοια. Θα πρέπει ο εθελοντισμός και ο ραστεχνισμός να ενταχθούν στον τομέα της δημιουργικότητας ώστε να ανακύψει μια πραγματική δημιουργική και αλληλέγγυα οικονομία. Η πρόσβαση στη δημιουργικότητα και στη γνώση αποτελούν ένα παράγοντα καθοριστικό όσον αφορά τα βασικά δικαιώματα, ιδιαίτερα για τα άτομα τα οποία είναι σε λιγότερο ευνοϊκή κατάσταση είτε λόγω κοινωνικής θέσης είτε λόγω προέλευσης φιλετικής ή εθνοτικής και η Ευρώπη. Η Ευρώπη σημαίνει κινητικότητα και ανταλλαγέ. Γι' αυτό ακριβώ θα επιθυμούσαμε να ενθαρρύνουμε πρωτοβουλίε όσον αφορά την κινητικότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά νέου που εκφράζουν την δημιουργικότητα και ζητάμε από τι χώρε μέλη να άρουν του φραγμού στην δημιουργικότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε χώρες εκτός Ευρώπης. Ζητάμε επίσης να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ της βιομηχανία, του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα στον τομέα της εκπαίδευση, της κατάρτιση και βεβαίως της ε, διαβίου μάθηση. Ιδιαίτερα στις ψηφιακές τεχνολογίες και στην αναγνώριση αυτών των δεξιοτήτων. Τέλος, θα ήθελα να επιμείνω για την ανάγκη διασφάλισης σε όλους τους εργαζομένους και ιδιαίτερα στους καλλιτέχνες, στους ανθρώπους του θεάματος, σε όλους τους δημιουργούς ότι η ευρωπαϊκή διαφορετικότητα θα πρέπει να τους διασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα όσον αφορά το επίδομα ανεργίας, την προστασία κατά των εργατικών ατυχημάτων, τα συνταξιωτικά τους δικαιώματα και μάλιστα, όπως είδαμε και την περασμένη εβδομάδα και το συζητήσαμε ε, στην Ολομέλεια, τα... τις άδειες πατρότητας και μητρότητας. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Μέχρι τις 10 του Νοέμβρη μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες και θα εισακούσω προσεκτικά τις δικές σας τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης. Μετά θα υιοθετήσουμε διακόπτη πρόεδρος. Θα σταματήσουμε εδώ, ε, κυρία Συγγήτρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δεχθώ λοιπόν προσεκτικά τις τροπολογίες σας. Θα πρέπει να διώσουμε του ρόλου μα, λέει η Πρόεδρος. Κυρία Στάνερουκ, Μπεναμιά. Στάνερουκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, κλάδη πολιτισμού και δημιουργικότητας είναι τομέας ανάπτυξης ε, το βλέπω και στη Γερμανία αυτό με τα στοιχεία που έχουμε και γι' αυτό πραγματικά είναι σωστό να έχουμε τώρα ένα σχετικό, μια σχετική πράσινη βίβλο. Και επίσης ε, είναι απαραίτητο να δούμε τις ε, κοινωνικές πτυχές και τις πτυχές απασχόλησης. Η πράσινη βίβλο της Κομισιόν, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ γενική και επί των αρχών και δεν αναφέρεται στις ε, στην κοινωνική πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συγχύτρια για την γνωμοδότησή της, γιατί περέλαβε πάρα πολλά στοιχεία που είναι σημαντικά για μας, κοινωνική ασφάλιση και η μείωση των διακρίσεων. Οι τροπολογίες μας θα αναφερθούν συγκεκριμένα στον τομέα αυτό, ασφάλιση διαβίωσης και την κοινωνική εξασφάλιση και μικρομεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, το θέμα της ε, χορήγησης κοινοτικών πόρων για τον τομέα της, ε, του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Λουκάς Μπεν Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και την εισηγήτρια. Ξέρω ότι δεν μπορεί κανείς να τα γράψει όλα για κάθε θέμα, αλλά θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο στο θέμα των δυνητικών θέσεων εργασίας. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για τη δημιουργία θέσεων στον καλλιτεχνικό τομέα και στις μικροεσαίες επιχειρήσεις παντού υπάρχουν θέματα, υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις των τεχνικών του θεάματος στα φωτιστικά, στον ήχο κτλ. Και έπειτα το είπε αλλά θέλω να επιμείνω ακόμη περισσότερο ελεύθερη κυκλοφορία ο αριθμός των καλλιτεχνών κάθε επίπεδο που μας μιλούν για την έλλειψη δυνατότητας μετακίνησης επειδή δεν παίρνουν βίζα. Δεν μιλάω βέβαια για τους καλλιτέχνες μέσα στην Ένωση, ας πούμε για τους Αφρικανούς καλλιτέχνες με τους οποίους ερχόμαστε σε συμφωνίες διαπραγματεύσεις. Πολλές φορές δεν μπορούν να έρθουν και να εκφραστούν στις χώρες μας, ιδιαίτερα στη Γαλλία, γιατί δεν έχουν θεώρηση. Ε, ενώ είναι φανερό ότι ειδικά στον καλλιτεχνικό τομέα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. Υπάρχει και η Ένωση για τη Μεσόγειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτές τους οργανισμούς πρέπει να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των καλλιτεχνών και όσων τους συνοδεύουν, των τεχνικών δηλαδή. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κώστα. Ναι, ευχαριστώ την εισηγήτρια και εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια στα πλαίσια της Επιτροπής Πολιτισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή μας αυτή να τονίζει εκτός από τις ε, κοινωνικές πτυχές αλλά και τις πτυχές που αφορούν τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και να υπάρχει μια μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική διάσταση του τρίτου τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Εδώ ακριβώς θα έπρεπε λοιπόν να κάνουμε και μία διευκρίνηση αναφερόμενη στο ψήφισμα που είχαμε για την κοινωνική οικονομία επειδή ο τομέας αυτός περιλαμβάνει πολλές μηχανίες και περιλαμβάνει πολλούς φορείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ιδρύματα, συνεταιρισμοί κλπ. κλπ. Οπότε το καθεστώς αυτό θα πρέπει να δούμε πιο προσεκτικά όσον αφορά και τους φορείς αλλά και κάποιους τομείς παραγωγής που δεν σχετίζονται απαραίτητα όσον αφορά με την καθαρή έννοια της βιομηχανίας. Μετά όσον αφορά την πτυχή της απασχόλησης είχαμε μία ακρόαση στη χώρα μου την Ιταλία με όλους τους φορείς αυτού του τομέα επειδή ω σκιώδη ήθελα να ακούσω τι διάφορε απόψει. Υπάρχει παραδείγματι ένα μεγάλο αίτημα για αναθεώρηση των τομέων που κάποιο θα είπε νομίζω νωρίτερα, τομέων όπως της μόδας, του πολιστικού τουρισμού, η βιομηχανία του γούστου όπως λέγεται στην Νότια Ευρώπη. Αυτοί οι τομείς λοιπόν σχετίζονται άμεσα με τον τομέα, με την βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργικότητα. Και εδώ έχουμε τομείς που ανέρχονται σε 8. Αυτός ο αριθμό μας φαίνεται περιοριστικό σε σχέση με, το, με το ευρύ σκηνικό που περιλαμβάνει αυτός ο τομέα και τους αντίστοιχου εργαζόμενους. Να υπενθυμίσω ότι στο τομέα του πολιτισμού και τη δημιουργικότητα, ένας από τους δύο εργαζόμενους είναι πτυχιούχος ή έχει σημαντικές δεξιότητε. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε μια σημαντική δυνατότητα καινοτομία, ποιοτική ποιοτικής Και νομίζω ότι υποεκτιμάμε στην πράσινη βίβλο την κληρονομιά των τοπίων και όλων των σχετικών τομέων. Οπότε θα πρέπει να δούμε ακριβώς και τις απαιτήσει που θα έχουμε εδώ και να έχουμε καλύτερη αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτήσει όσον αφορά τις δεξιότητες στον τομέα αυτό, που περιλαμβάνει σημαντικές διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες. Και δύο τελευταία πράγματα ακόμα. Συμφωνώ με αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως όσον αφορά το θέμα της κινητικότητας των καλλιτεχνών όσον αφορά εξάλλου και τη δέσμευση για το έτος της Ευρωπαϊκής Δημιουργικότητας και Πολιτισμού που δεν, είχαν και τόσο, που είχε και τόσες επιπτώσεις για να κάνουμε ακριβώς πιο εύκολη την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των πολιτιστικών φορέων. Ε, για το θέμα αυτό να πω ότι παρόλο που το συζητήσαμε στην Επιτροπή Πολιτισμού να πω ότι οι εκδότες πρότειναν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι εκδότες δηλαδή να προβλέψουμε ένα πρόγραμμα Media το οποίο αφορά σήμερα μόνο τα οπτικοακουστικά να έχουμε ένα κομμάτι του Media το οποίο θα υποστηρίζει και τις ανεξάρτητες ε, τους ανεξάρτητους εκδοτικούς οίκους που κάνουν ε, μεταφράσεις έργων λιγότερα γνωστών στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν, να έχουμε λοιπόν και κάτι αντίστοιχο για αυτό το τομέα. Τελευταίο ζήτημα πνευματικά δικαιώματα. Ξέρουμε ότι τα πνευματικά δικαιώματα είναι κάτι το οποίο ήταν αντικείμενο ψηφίσματος. Όμως οι αμοιβέ των φορέων δημιουργικότητας θα πρέπει να τονιστεί εδώ γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης της ανέχειας ώστε να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ πραγματικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των δημιουργών. Γιατί αναφέραμε ε, προηγουμένως ότι στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας η, η θέση εργασίας δεν είναι και τόσο ασφαλής, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την κοινωνική πρόνοια όσον αφορά αυτούς τους ε, φορείς πολιτισμού και δημιουργικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Μάρκινγκ και Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Σκιώδη μου έστειλε κάποιε σημειώσει γιατί δεν μπορούσε να έρθει σήμερα το απόγευμα εδώ, να πω κάποια πράγματα εκ μέρου του. Κατά λοιπόν θα ήθελε να ευχαριστήσει την εισηγήτρια, αλλά θα ήθελε να κάνει κάποιε προσθέσει. Προσθήκη, συγγνώμη. Θα ήθελε να δοθεί περισσότερη ε, έφαση σε κάποια θέματα και να γίνουν κάποιες αλλαγές. Ε, οι λεπτομερείς ε, προτάσει αφορούν τα εξή. Στην παράγραφο 1, βεβαίω συμφωνεί με την κλίση προ τι χώρε μέλη για να θεσπίσουν αλλαγή όσον αφορά τα συστήματα κοινωνική πρόνοια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκε των δημιουργών όσον αφορά το τομέα του πολιτισμού και τη μερικότητα. Όμω, τα κοινωνικά συστήματα στου τομεί αυτού θα πρέπει να είναι ευέλικτα, επειδή η ευελιξία είναι τους, η λέξη κλειδί, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είτε είναι ε, ανεξάρτητοι, είτε μη ανεξα... απασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι ή μη αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι πολύ συχνά αντιμετωπίζουν άτυπη εργασία και σημαντικές περιόδους ανεργίας. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε φραγμό όσον αφορά τη δημιουργικότητα στον τομέα αυτό και θα πρέπει η κοινωνική πρόνοια να είναι ίση για όλους τους συμμετέχοντες σε οποιοδήποτε τομέα. Επίση, τονίζει το γεγονό ότι το CCI, ένας πολύς, η βιομηχανία αυτή είναι πάρα πολύ οικονομικός τομέας επειδή έχει και παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές προοπτικές. Τονίζει λοιπόν την σημασία του τομέα αυτού ως οικονομικού τομέα και Τονίζει επίσης την σημασία του όσον αφορά την δημιουργία, την προοπτική δημιουργίας θέσεων εργασίας. Επίσης αναφέρει το γεγονό ότι η βιομηχανία του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αφορούν την διαχείριση, την επιχειρηματική επίσης, οπότε τα άτομα αυτά δεν θα πρέπει να α, μην έχουν τα απαραίτητα πτυχία, τι απαραίτητε δεξιότητε και τι οικονομικέ αυτή την περίπτωση. Οπότε αυτέ θα πρέπει να διαθέσουμε σε όλου. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε τη σημασία τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση όσον αφορά του φορεί πολιτισμού και δημιουργικότητα. Και το τελευταίο που θα ήθελα να τονίσει είναι το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων. Κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη απειλή για το τομέα αυτό. Θα πρέπει να δούμε ε, Κάποιε λύσεις, κάποιε δυνατότητες, όπως κάποιο πρόσθετο φόρος που έχει εφαρμοστεί σε κάποιε χώρε όπως το Βέλγιο. Να προσθέσω και εγώ τα δικά μου σχόλια. Πιστεύω θα πρέπει να δούμε ποια είναι ακριβώ τα διακυβευόμενα και θα πρέπει να σχετίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα με τη στρατηγική 2020 όσον αφορά την καινοτομία και την ε, ψηφιακή ατζέντα, νέε θέσει εργασία, νέε δεξιότητε κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Μπαλτισά μετά η κυρία Αλήν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την συγκήτρια για τη θαυμάσια εργασία που έκανε. Στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης ακούσαμε την άποψη ενός εμπειρογνώμονα για την καταπολέμηση τη ανεργία, για το πώ θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασία σε αυτή την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα από του τομεί που ομόφωνα καταδεικνύεται ω τομέα που παρουσιάζει μεγάλε δυνατότητε για την δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασία που φαίνεται σήμερα να λείπουν από, τον, από την Ήπειρό μα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιλάβουμε κάποιο πιο έτσι έντονο και εμφαντικό στοιχείο εδώ, γιατί νομίζω ότι στην νομοδότηση γίνεται σαφής αναφορά στις στρατηγικές για την ενίσχυση και συγκεκριμενοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης του τομέα αυτού. Αναφέρεται το θέμα το, της ψηφιακής ανάπτυξης, της ευρωπαϊκής ατζέντα, η διεύρυνση της ψηφικοποίησης ψηφιοποίηση στο ευρωπαϊκό σύστημα, θέματα τα οποία επαναλαμβάνονται και εμφανίζονται σε διάφορα έγγραφα, θα πρέπει όμω να είμαστε συγκεκριμένοι για το πώ ακριβώ θα θέλαμε να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Όπω επίση και η ένωση καινοτομία που θα πρέπει να κάνουμε, δηλαδή αυτή η ανάγκη παρέμβαση και οικονομική υποστήριξη των τομέων του πολιτισμού και της γεωργικότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν συγκεκριμένα εργαλεία γιατί ο τομέας είναι ιδιάζοντας. Υπάρχει ένας τομέας όπου υπάρχει υψηλό ποσοστό τεχνολογίας, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπάρχουν άλλοι τομείς όπου δεν έχουμε άμεσα αποτελέσματα αλλά θα πρέπει να συνοδεύουμε τους τομείς αυτούς με κάποια εργαλεία τα οποία θα πρέπει να είναι ιδιάζοντα για τον κάθε τομέα και νομίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και αυτό που είπαν και οι προλαλήσαντες το, σημείο δηλαδή της στρατηγικής προσέγγισης για το πώς θα πετύχουμε αυτή την ισορροπία, αυτόν τον συμβασμό μεταξύ πνευματικών δικαιωμάτων και Τη προώθηση νέων μορφών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα έχει σημασία το θέμα που αφορά την κοινωνική πρόνοια των εργαζομένων στον τομέα αυτό, επειδή ακριβώς τα χαρακτηριστικά κάποιων τομέων του πολιτισμού και της ε, δημιουργικότητας αντιμετωπίζουν αυτή την έλλειψη συνεχούς εργασίας, κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την κατάσταση όσον αφορά την συνταξιοδότηση, την μελλοντική των εργαζομένων στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Yes, thank you. Uh, just a couple of remarks. Σας ευχαριστώ λίγα σχόλια μόνο. Αναφέρθηκατε στι αλλαγές στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των πρώτων μελών. Πώς φαντάζεστε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί προφανώ η κοινωνική ασφάλεια δεν είναι δική μα αρμοδιότητα. Η τρίτη παράγραφο αναφέρεται στην ελεύθερη κυκλοφορία, ιδίω σχετικά με τι ανταλλαγέ μεταξύ καλλιτεχνών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ χωρών τη ΕΕ και τρίτων χωρών. Εμεί δεν είμαστε αρμόδιοι για το θέματα μεταξύ χωρών τη ΕΕ και τρίτων χωρών. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό της ΕΕ. δεν θα μπορέσουμε να δούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν θα πρέπει γι' αυτό ίσω να αναφερθούμε στι χώρε, στι τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναφερθούμε στην ελεύθερη κυκλοφορία μεταξύ των χωρών τη ΕΕ. Εκτό είναι δύσκολο να αναφερθούμε. Πρόεδρο, άλλο θέλει το λόγο. Δεν βλέπω, θα κάνω και εγώ κάποιε παρατηρήσει. Η πρώτη είναι ότι η ανακοίνωση τη Κομισιόν αναφέρεται στους κλάδους πολιτισμού και δημιουργικότητας. Είμαστε λοιπόν εδώ σε μια στρατηγική, ε, αν θέλετε, που θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα της βιομηχανικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όσον αφορά τις αρμοδιότητες δικής μας επιτροπής, το πρώτο θέμα είναι η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων απασχόλησης από τον κλάδους αυτούς. Ελπίζω να έχουμε ένα συμβασμό για να φανεί αυτό το θέμα πρώτο πριν να αναφερθούμε στις Το ανέφεραν οι διάφοροι ομιλητέ αυτό. Τώρα δεν ξέρω πού θα οδηγηθεί αυτή η ανακοίνωση Κομισιόν. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα δυναμικό που δεν έχει τύχει πλήρως εκμετάλλευσης ε, και κατά κάποιο τρόπο αυτό σχετίζεται με την αξιολόγηση εκεί, των ταλένων εκείνων των ε, πολιτών που βρίσκονται κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά που λέμε για την έξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την κρίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε το δυναμικό της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Η καινοτομία, η δημιουργικότητα θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο πολλαπλασιαστή, πάρα πολύ σημαντικό για την απασχόληση. Και αυτό είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Υπάρχουν κάποιες ιστορίες επιτυχίας στην Ευρώπη σχετικά το παρελθόν, γιατί να μην ξαναγίνει σήμερα. σκέπτομαι τα Λέγκο παραδείγματο χάρη. Υπάρχουν και άλλες όμως. Που ξεκινούν από μια ιδέα και από εκεί αναπτύσσεται μια τεράστια βιομηχανία. Πολύ παραγωγική. Όσον αφορά τους κοινωνικές προϋποθέσεις υπάρχουν διάφοροι παράγραφοι πολύ ενδιαφέρουσες όσον αφορά συμβολή μας στο κείμενο αυτό. Θα πρέπει να ξεχνάμε και τις εργασίες ε, κατά τα άλλα τη Επιτροπής μας. Ξέρω βέβαια ότι δεν έχουμε πολλές δυνατότητες να αναπτύξουμε το θέμα στην περίπτωση αυτή. Αλλά για τα κοινωνικά, ίσως είμαστε υπερβολικά περιορισμένοι. Γιατί πριν μπούμε στις λεπτομέρειες των συστημάτων κοινωνικής προστασίας κλπ. κλπ υπάρχει κάτι πολύ πιο σφαιρικό. Δηλαδή θέλουμε την ανάπτυξη των θέσεων αυτών απασχόλησης και του δυναμικού απασχόλησης που προσωπεύει η βιομηχανία αυτή. Από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι πρόκειται για βιομηχανίε όπου η τάση για άτυπες μορφέ εργασία μπορούσε να ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και όλα αυτά που λέμε κατά τα άλλα για τις άτυπες μορφέ εργασία και τους όρους εργασία και κοινωνική προστασία, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και εδώ. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό που εξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα και αυτή την πρωτοβουλία της Κομισιόν και φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα πρόγραμμα πιλότο και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τον δανεισμό που υπάρχει νομίζω εδώ. Εάν δεν θέλει κανένα άλλο να θέλει το λόγο. Α, η κυρία Μαρά. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε γιατί ήρθα καθυστερημένη στη συνεδρίαση, αλλά άκουσα την ανάλυση σας, συμφωνώ με πολλά από όσα είπατε, καταρχήν για την αστάθεια αυτών των θέσεων στον τομέα των νέων τεχνολογιών, είναι θέσεις πολύ πτυτικές. Δεν διαρκούν πολύ χρόνο. και πρόκειται για προσλήψεις πάνω σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και που περιορίζονται σε αυτό. Πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι εδώ αλλάζει το γνωστό σχήμα εργασίας και πρόσληψης. Δεύτερον, και πρέπει να το πούμε και ως προς το 3 και 4, σε όλες αυτές τις καινούργιες θέσεις στον τομέα της παραγωγής υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ τελείως διαφορετικών δεξιοτήτων δηλαδή πρόκειται για δεξιότητες δημιουργίας και σύλληψης από τη μία και από την άλλη καλλιτεχνικής ενίσχυσης του σχεδίου Αυτό θα ήθελα να φαίνεται πιο πολύ καλύτερα στο κείμενό μας γιατί αν παραμείνουμε στο κείμενο που έχουμε τότε θα παραμείνουμε στα λεγόμενα νέα μέσα πρόσληψης του πολιτισμού. Ενώ εδώ πρόκειται για κάτι το τελείως διαφορετικό. Για νέα σύλληψη της μαθητείας με βάση αυτά τα νέα επικοινωνιακά μέσα. Αυτά είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα πρότυπα, γιατί δεν υπάρχουν ακόμη και πρέπει να δημιουργηθούν τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να φαίνεται καλά το τμήμα της δημιουργίας από τη μία και της σύλληψης από την άλλη. Αυτή είναι και η διαφορά μεταξύ της παιχνιδιάρικης μαθητείας και της κλασικής. Αγαπητοί συνάδελφοι και κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή της γνωμοδότησης. Όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά κυρία Πρόεδρε, είμαστε, έχουμε πίεση χρόνου και δεν μπορούμε να τα γράψουμε και όλα, αλλά νομίζω ότι ένας από τους κύριους και πραγματικούς άξονες είναι ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας θέλουμε να αφορά την ποιοτική εργασία και το πρόβλημα με τις τρίτες χώρες, τις τρίτες χώρες και πρέπει να το ξαναδούμε αυτό είναι, για να είναι τα πράγματα πιο σαφή είναι ότι πρέπει να τονίσουμε την κινητικότητα ως προς τις ανθρώπους που προέρχονται από τρίτες χώρες, το είπε και ο κύριος Μπεναχμίας. Αλλά πάντως ε, αυτά, αυτές οι προσθήκες ε, είναι ευπρόσδεκτες από μένα στην ορμαδότησή μου. Τελείωσε η συζήτηση. Χρονοδιάγραμμα. Το είπε και η συγγήτρια. Αρμόδια Επιτροπή 25 Ιανουαρίου διορία κατάδειξη των προγειων 25 25-26 Οκτωβρίου του Αγίου Δημητρίου. Όχι, 10 Νοεμβρίου. 10 Νοεμβρίου το μεσημέρι. Έτσι ώστε να έχουν μεταφραστεί κατά την εξέτασή μας την 1η Δεκεμβρίου και να τις ψηφίσουμε την, στις 2 Δεκεμβρίου. Έληξε η σημερινή μας συνειδρίαση. καλή και θα τα ξαναπούμε αύριο στις 9 με τις κάρτες σας όμως. Με τις κάρτες.